Okay, um, Ας αρχίσουμε λοιπόν για την ε, κοινοβουλευτική εποπτεία. Είναι η τρίτη ενότητα. Η κοινοβουλευτική εποπτεία των υπηρεσιών, ε, ε, των μυστικών υπηρεσιών. Καλωσορίζω τον κύριο Ιεν Κάμερον της Επιτροπής Βενετίας που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του νόμου. Είναι επίσης καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Και το κείμενο ε, της ομιλίας του θα μας το διανύμει σε όλους μετά τη λήξη της παρουσίασης. Έχετε το λόγο, Ιέν. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε χωρίς μικρόφωνο. Sorry, uh, I will speak a little. Συγγνώμη. Να σας πω λίγο ποια είναι η έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας για το 2007 για τη δημοκρατική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας. Ε, χρειάζεται κάποια ενημέρωση αυτή η έκθεση. Εγώ είμαι συγγητής και η ενημέρωση θα συζητηθεί και ελπίζω να εγκριθεί και από την Ολομέλεια Μάρτιο συγγνώμη, του 2014 στην Επιτροπή της Βενετίας. Ποιοι είναι μέλη εκεί. Ίσως γνωρίζετε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των διαφόρων επιτροπών με 25 ετή και πλέον εμπειρία για θέματα συνταγματικά διεθνούς δικαίου και ε, γνωρίζουν πολύ καλά πώς λειτουργεί η κατάσταση, έχουν τεράστια εμπειρία για τους μηχανισμούς ε, πολιτικής λογοδοσίας και ε, εποπτείας. Επιτρέψτε μου να σας πω και μερικά πράγματα για τα ειδικά προβλήματα ε, εποπτείας της στρατηγικής παρακολούθησης. Η έκθεση είναι 60 σελίδων, έκθεση του 2007 της Επιτροπής Βενετίας και εξετάζει μοντέλα και τρόπους λογοδοσίας έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες και τα δυνατά σημεία αυτών των μεθόδων και επηρέασε πάρα πολύ τις επόμενες εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρομοκρατία, ε, καθώς επίσης και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2011 που ακολούθησε. Η έκθεση του 2007 δεν εξετάζει συγκεκριμένα και ειδικά τη στρατηγική παρακολούθηση, αλλά η ενημέρωση, η νέα έκδοση θα ασχοληθεί με αυτό στο βαθμό που έχει επιπτώσεις και στην εσωτερική ασφάλεια. Να πω κάτι για το πρόβλημα. Μπορούμε πολύ απλά να το περιγράψουμε ως εξής. Οι ε, δημοκρατικές κοινωνίες είναι βάλωτες και ταυτόχρονα ε, είναι και συγκεχημένη η φύση των απειλών ε. Δηλαδή σήμερα το χρησιμοποιούν αυτό για οποιοδήποτε λόγο και μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο. Αν δεν τεθούν λοιπόν εξωτερικά όρια και περιορισμοί, τα οποία θα επαναλαμβάνονται συνέχεια, η φυσική τάση που έχουν όλες οι μυστικές υπηρεσίες και πληροφοριών θα είναι να συλλέγουν υπερβολικές πληροφορίες. Και αυτό φαίνεται ε, από την παρούσα έρευνα πολύ εύγλωτα. Ε, τα εσωτερικά όρια δεν πρόκειται να είναι αρκετά ούτε ικανοποιητικά. Για ποιο λόγο το προσωπικό των υπηρεσιών αυτό να αυτοπεριορίζεται σε ένα δημοκρατικό κράτος δεν είναι βασικά και η δουλειά τους στο κάτω-κάτω. Να σκεφτούν τι συνέπειες και τι βλάβες και ζημίες μπορούν να προκαλέσουν σε μια δημοκρατική κοινωνία όταν συλλέγουν υπερβολικές πληροφορίες. Και θα γνωρίζετε τώρα ότι οι κασίες και καταγγελίες που εξετάζονται από την έρευνα αυτή αφορούν κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένε Πολιτείες που είναι και οι δύο δημοκρατικές χώρες. Και τελικά οι δημοκρατικά εκλεγμένοι ε, πολιτικοί θα πρέπει ε, να είναι οι φυσικοί ελεγκτές ε, ας πούμε των μυστικών αυτών υπηρεσιών. Όπως γνωρίζετε ο φυσικός και ο διοικητικός έλεγχος και οι δυνατότητες ε, στο παρελθόν έχουν θέσει ε, κάποια όρια και πόσο μπορεί κανείς να επεμβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο μεταξύ όμως η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια πρόοδο για τη συλλογή, ε, αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και έτσι έχει αυξηθεί δραματικά η δυνατότητα των ε, μυστικών αυτών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας. Και πάλι πολύ εύγλωτα το περιγράφει αυτό η παρούσα έρευνα. Και το θέμα δεν είναι μόνο να συλλέγονται στοιχεία. Τα μαζεύουν για να τα χρησιμοποιήσουν με διάφορους τρόπους. Σε ε, ε ποινικέ έρευνες ε, για να έχουμε πιο στοχευμένες κυρώσεις, έλεγχο ασφαλείας για αποφάσεις σχετικές με τη χορήγηση ηθαγένειας ή απέλασης αλλοδαπών και βεβαίως ε, το πιο επίμαχο είναι για εξωτερικά θέματα, ε, επιθέσεις με ε, μη επανδρομένα σκάφη ή παραδόσεις, renditions. Τέσσερα είναι λοιπόν τα είδη της λογοδοσίας προς το κράτος, πέρα από την εσωτερική. Και αυτές είναι κοινοβουλευτική, δικαστική, σε ανεξάρτητες αρχές εμπειρογνωμόνων και ε, ε, μηχανισμοί καταγγελιών. Τα δύο τελευταία είναι μηχανισμοί ε, υποκατάστασης ή αντικατάστασης των δύο πρώτων των κοινοβουλίων και των δικαστηρίων που δεν λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα γνωρίζετε λοιπόν ότι από τη φύση τους οι μυστικές αυτές υπηρεσίες σε μεγάλο βαθμό στόχο έχουν την εκτίμηση κινδύνου και ρίσκου. Και αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί λογοδοσίας, για να υπάρχει και μια δεύτερη γνώμη ουσιαστική ε, για αυτά τα θέματα, δεν υπάρχουν πραγματικά εχέγγυα. Και στη χειρότερη περίπτωση μπορείτε να έχετε μηχανισμούς που αυτονομούνται και δεν είναι καθόλου ε, ασφαλιστικές δικλείδες παρά μόνο ιδεολογικά ε, προπετάσματα καπνού. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε λοιπόν εξωτερική έλεγχη με βασική αποστολή την υποστήριξη ή την ενίσχυση των εσωτερικών ε, υφισταμένων ελέγχων. Το προσωπικό ναι. των μυστικών υπηρεσιών υπηρεσιών ασφαλείας είναι προσιλωμένο στις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η πρώτη εγγύηση. Ναι η Επιτροπή της Βενετίας δεν αποφέρεται αν θα πρέπει η υποπτία να είναι ε, κοινοβουλευτική από πλευράς ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων ανάλογα με τη χώρα μπορεί να υιοθετηθεί διαφορετικό σύστημα ε, και ανάλογα με τη συνταγματική τάξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν και τα δύο. Και κοινοβουλευτική εποπτεία και από εμπειρογνώμονες. Βέβαια, οι βρυδικές μορφές δεν ξέρω αν μπορούν να υπάρξουν. Οι σκανδιναβικές χώρες το έχουν, Νορβηγία, Σουηδία σε ό,τι αφορά την στρατηγική εποπτεία και επισκόπηση, τα αμυγό κοινοβουλευτικά συστήματα δεν λειτουργούν, δεν αποδίδουν. Καλό θα ήταν να γνωρίζουμε εδώ ότι υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που απαιτεί ε, ε, ανεξαρτήτους ελέγχους και κατά την έγκριση ε, και κατά την διαξαγωγή της έρευνας και της συλλογής. Στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν διαπιστώσει Ε, ότι βεβαίως υπάρχει το δικαστήριο FIAC, αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται ένα σύστημα ε, συνέχειας και παρακολούθησης αυτού του θέματος που ε, χρειάζεται ένα εξωτερικό σώμα εμπειρογνωμόνων και ανεξάρτητο με ίδιες ερευνητικές εξουσίες. Υποθέτω ότι σήμερα το πρωί συζητήσατε την έκθεση αυτή και συμφωνώ με μερικά από τα συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω είναι λάθος να ανακατεύονται οι διάφοροι εθνικοί μηχανισμοί επισκόπησης, πράγμα που κάνει η μελέτη. Το βρετανικό σύστημα είναι κατακαιρματισμένο και ακατάλληλο για την επισκόπηση και εποπτεία ως προς τη στρατηγική παρακολούθηση. Ενώ το γερμανικό και το σουηδικό σύστημα δεν είναι καθόλου κακά. Δεν λέω ότι δεν χωρούν βελτιώσεις, αλλά καλούτσικα είναι. Ε, υπάρχει έλεγχος πραγματικά θεσμικός και ορίζεται σαφώς τι μπορεί να κάνει η υπηρεσία και τι δεν μπορεί να κάνει με μικρές ε, επιχειρήσεις σε αντίθεση, σε σύγκριση με τους ε, ε αγγλικούς και αμερικανικούς μηχανισμούς και είναι πολύ ισχυρότερο ο έλεγχος. Λοιπόν, να σας αναφέρω τελειώνοντας τρία βασικά προβλήματα προς τη στρατηγική παρακολούθηση. Το πρώτο, η εποπτεία και η επισκόπωση αυτή. προβλήματα υπάρχουν και λύσεις υπάρχουν και πολλές χώρες μπορούν να τις ε, αποδείξουν στην πράξη και να υιοθετήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Πρώτον, πολύ αρνητικέ επιπτώσεις της μαζικής παρακολούθησης στην ε, κοινωνία δεν χρειάζεται να τις εξηγήσω. Μια προφανής λύση είναι να ε, περιοριστεί η συλλογή όσο γίνεται, οι πηγές. Δηλαδή, να ορίζεται σαφώς τι επιτρέπεται να συλλέγουν ως στοιχεία οι υπηρεσίες και τι δεν θα πρέπει να συλλέγουν. Και η γερμανική και η σουηδική νομοθεσία αποτελούν εδώ χρήσιμα μοντέλα προς μίμηση. Ένα δεύτερο όριο που μπορείτε να βάλετε είναι να περιοριστεί η χωρητικότητα, η δυνατότητα ε, συλλογής ε, μια χρονική μονάδα. Και πάλι το γερμανικό παράδειγμα είναι εδώ καλό και εξ όσων γνωρίζω περιορίζεται στο 20% μια ε, χρονική στιγμή δεδομένη. Τρίτον, να ε, απαγορεύονται οι μαζικές μεταφορές χίδιν ε, στοιχείων, bulk data. Τέταρτο, μπορεί να απαγορεύεται επίσης η συλλογή τέτοιων στοιχείων για εμπορικούς σκοπούς και να μην ασχολείται το Υπουργείο Εμπορίου με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν τρεις τομείς τουλάχιστον επαγγελματικών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμπορικών που είναι πολύ χρήσιμο και ε, θεμητό να ελέγχεται η δραστηριότητα. Το πρώτο είναι τα ε, όπλα μαζικής καταστροφής και η διάδοσή τους, ε, η ψυχία διτής χρήσης, εξαγωγή. Όταν είσαι μια οικονομία σαν τη Γερμανία εξαγωγικής ε, φύσεως, καλό είναι να κοιτάς που πηγαίνουν αυτά τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για ειρηνικούς και για πολεμικούς σκοπούς. Άλλο στοιχείο είναι το, η μαζική ε, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα δηλαδή και ε, επίσης οι τηλεπικοινωνίες και το εμπάργο. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που επίσης μπορεί να λυθεί είναι το ρίσκο, ο κίνδυνος να υπάρχουν σφάλματα. Όταν αναμειγνύονται ε, βάσεις ιδιωτικών προσωπικών δεδομένων με δημόσιες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει ξανακοιτάξει αυτό το θέμα. Ε, στο PNR τα ε, στοιχεία των επιβατών αεροπορικών πτήσεων και ε, άλλα. Αυτό είναι το data mining και είναι πολύ σημαντικό αυτό το φακέλωμα. Μπορεί να υπάρχουν ιδιωτικοί μεμονωμένοι φάκελοι, αλλά με ανώτατα όρια. Και θα πρέπει να γίνεται σωστή επεξεργασία και παρακολούθηση των στοιχείων αυτών που συλλέγονται από ιδιώτες με σωστή σήμανση και ο ε, οργανισμός που ελέγχει και εποπτεύει θα πρέπει να έχει ειδική ε, δυνατότητα να ε, ελέγχει τα προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως εθνικότητας. Και το τελευταίο, υπάρχει δυνατότητα στη στρατηγική παρακολούθηση να χρησιμοποιείται αυτή για να παρακάμπτονται πιο αυστηροί εθνικοί έλεγχοι για λόγους επιβολής του νόμου από τις διοκτικές αρχές. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τα τηλεφωνήματα, οι επικοινωνίες εντός μιας χώρας μπορούν να παγιδευτούν ε, από κάποιο διεθνή παράγοντα. Και ένα τοπικό τηλεφώνημα γίνεται πολύ γρήγορα διεθνές. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά, ότι ε, ορισμένες ε, εταιρείες και μυστικές υπηρεσίες κατασκοπεύουν ε, τους πολίτες ο ένας το άλλο προς λογαριασμό της τρίτης υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να απαγορευτεί. Δεν μπορείς να ζητήσεις από μια μυστική υπηρεσία να παρακολουθεί τους πολίτες όταν απαγορεύεται να το κάνεις εσύ. Αλλά αυτό που δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει είναι η παθητική ε, λήψη στοιχείων από άλλες υπηρεσίες. Ναι, πού θα τραβήξει εκεί τη διαχωριστική γραμμή θα ήταν ε, άστοχο να ε, απαγορευτεί οποιαδήποτε παθητική λήψη στοιχείων. Δηλαδή όταν θέλει να σε ειδοποιήσει μια άλλη μυστική υπηρεσία για κάτι που πάει στραβά θα πεις «Α, όχι, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το στοιχείο». Όταν γίνονται υποκλοπές, ας πούμε, οι παγιδεύσει τηλεφώνων και σου θέτουν υπόψη ότι κοίτα πρέπει να το κοιτάξεις, δεν μπορείς να πεις ότι «Α, όχι, δεν επιτρέπεται». Αυτό και πάλι μπορεί να έχει μερική μόνο κάλυψη. Γιατί ξέρετε ότι ε, θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους ε, ε, στην επικράτειά τους οι μυστικές υπηρεσίες μια χώρα. Και μάλιστα μπορεί κανείς να δει από διάφορες νομοθεσίες. Η Γερμανία προβλέπεται κοινοποίηση και όταν η παρακολούθηση γίνεται ιδιαίτερα στοχευμένη και προσωπική, με κάποιες εξαιρέσεις, βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, ε, δίνεται λόγο στο υποπτικό όργανο, εάν ε, πραγματικά πρόκειται για εξαίρεση και θα πρέπει να εφαρμοστεί ή όχι. Και αυτός ο εποπτικός φορέας θα ε, μπορεί να διαβιβάζει σε αρμόδιες αρχές ε, πληροφορίες για πάρα πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και πάρα πολύ σοβαρές παραβιάσεις για να ε, ξεπεραστεί ο κίνδυνος της παράκαμψης ή του βραχικυκλώματος ως προς τις ξένες υπηρεσίες. Γενικά λοιπόν οι εποπτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν θα πρέπει να έχουν ισχυρή εντολή όσο και ευρεία για να καλύπτουν όλα τα στοιχεία ε, ε, ε, της στρατηγική παρακολούθησης. Τέλος, συγκεκριμένη πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να αποφασίσει το Κοινοβούλιο για την ομοθεσία ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορεί να ενθαρρύνει καλές πρακτικές και να δημοσιεύει τις κακές και καλό θα ήταν να το πράττει κιόλα. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να βοηθήσει το υφιστάμενο δίκτυο των εποπτικών ε, αρχών στα κράτη-μέλη, στην Νορβηγία και την Ελβετία. Υπάρχει τέτοια συνεργασία, συνεδριάζουν τακτικά, αλλά το πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Είναι πολύ απλό είναι χρήσιμο το δίκτυο αυτό, η παραλαμβάνω έχει τακτικές συνεδριάσεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες, όχι απόρριτες, ε, ούτε εμπιστευτικέ, αλλά για κοινά προβλήματα, πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα με επαφέ τα προβλήματά τους. Εκεί μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο με ένα πολύ μικρό κονδύλι ε, και μπορεί να ενθαρρύνει αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Τίποτα, κύριε Κάμερον μου. Μήπως οι συνάδελφοι έχουν καμία σύντομη ερώτηση. Γιάννη θέλεις να αρχίσεις από τους σκιώδεις. Είναι οι σκιώδεις μας ξέρετε αυτοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάμερον για την παρουσία σας και για την πληροφόρηση που μας δώσατε για το πολύ σημαντικό θέμα των σχέσεων δημοκρατίας και εφταξίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αυτά τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης και η διαχείριση, η εκπαιρέωση που γίνεται των πληροφοριών που συλλέγονται δεν διαφοροποιεί τελικά την πληροφόρηση διαφορετικού τύπου που υπάρχει διαφόρων κατηγοριών. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της σχέσης δικηγόρου και πελάτη και πώς να υπάρξει προστασία των εσωτερικών συζητήσεων ενός κοινοβουλίου και εμπιστευτικός χαρακτήρας μεταξύ ιατρού και ασθενούς. Πώς. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, αλλά σύντομα. Τα λόμπι έχουν αυτοματοποιημένα συστήματα για αυτά τα πράγματα. Αλλά βασικά, καταρχάς πρέπει το προσωπικό να είναι καλά εκπεπεδευμένο να είναι αφοσιωμένο στις δημοκρατικές αξίες αλλά και πολύ σοβαρή εποπτεία. Όταν γίνουν όλα αυτά ατομικά χάνονται, χάνεται η προστασία. Το θέμα είναι όχι τα άτομα αλλά αν φτάσουμε μέχρι τα άτομα τότε πρέπει να υπάρχουν στεναρές εσωτερικές διαδικασίες για να επιτρέπεται τέτοια προσέγγιση με ατομική, σε ατομική βάση των λόμπι και να προσέχουμε την κάθε περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτε παραπάνω ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή περίπτωση με την περίπτωση άμα φτάσουν τα πράγματα ως το ατομικό επίπεδο. Κύριε Κόρνι Ένστ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Μισό λεπτό να βάλει κανένα ακουστικό. Τα γερμανικά μου είναι πολύ φτωχά. Also der Rechtsstaat äh, und die Το κράτος δικαίου και η απόρριτη δημοκρατία ε, δεν μπορεί να συμβαδίζουν πια. Ε, δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοιες δυσκολίες πλέον με αυτή τη μυστική διπλωματία, όταν μυστικές υπηρεσίες, πώς να το πω, έχουν όλο και περισσότερες κρίσιμες πληροφορίες. Αυτό είναι πρόβλημα για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και το βλέπουμε στην Επιτροπή μας, ακούμε όλο και περισσότερο ότι «Αχ, αυτό είναι απόρριτο, εμπιστευτικό και κλεισμένο των θυρών, αποκλείεται, άστο κάτω το χαρτί, δεν μπορείς να το πάρεις». Ε, και όλο και περισσότερες δυσκολίες. Για μένα είναι πρόβλημα αυτό για να ασκήσουμε τον έλεγχο. Και όπως εσείς ε, συμφωνώ, ε, είμαι ευνοϊκή και ε, προς ε, τον έλεγχο των εμπειρογνωμόνων γιατί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν αρκεί σε καμία περίπτωση. Και ιδιαίτερα για αυτά τα θέματα του απορρίτου και τα εμπιστευτικά μπορείτε να μας πείτε κάτι. Μπορούμε να συστήσουμε όσα όργανα θέλουμε. Αλλά αν δεν έχουμε δικαίωμα να βλέπουμε ε, χωρίς καμία ε, επιφύλαξη περιορισμό τα έγγραφα, αν δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη διάθεσή μας οι βουλευτές, ε, ας βάλουμε και λουκέτο, κατεβάσουμε τα ρολά. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό πια. Well, Συμφωνώ. Ο φορέα εποπτεία που θα υπάρχει θα πρέπει να είναι ένα φορέα που να αποτελείται από ειδικού και να έχει άμεση σχέση με το κοινοβούλιο. Διότι το κοινοβούλιο είναι αυτό που παρέχει την νομιμότητα προκειμένου να γίνουν όλα αυτά. Σωστά μιλάτε για ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, το κάτω-κάτω τη γραφή. Επίσης, χρειάζεται η νομιμότητα του Κοινοβουλίου με τακτικές επαφές και συνομιλίες με τους βουλευτές. Ακόμη και αν οι πλέον απόρριτες πληροφορίες δεν μπορούν να αποκαλύπτονται. Όμως, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να τους εμπιστεύεται και το κοινό... Οι πολίτε να εμπιστεύονται το κοινοβούλιο με τη σειρά του. Ένα πρόβλημα πρόσβαση στον τομέα αυτό είναι ότι δεν μπορούν να αποκαλυφθούν όλε οι πληροφορίε που έχουν μεταφερθεί από ξένου φορεί. Αυτός είναι ένας κανόνας για τις μυστικές υπηρεσίες. Μόνον το υλικό που μεταφέρεται μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών μπορεί να, δεν μπορεί μάλλον να αποκαλυφθεί σε καμία περίπτωση σε άλλους. Ο Εθνικός Εποπτικός Φορέας έχει δικαίωμα να δει αυτές τις πληροφορίες. Μόνον αυτός. Πρέπει να είναι σαφέσιμος αυτό στην ε, εντολή στην εντολή του φορέα εποπτείας. Βεβαίως, κάποιες πληροφορίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Υπάρχουν ε, καθαροτερημένες διαδικασίες για να τις χειριστεί κανείς, αλλά ο εθνικός εποπτικός φορέας μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες, ακόμα και αυτές που έχουν μεταφερθεί διοπηρεσιακώς, από ξένες ε, υπηρεσίε. Ευχαριστούμε, κυρία Σίπολ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η μαζική συλλογή δεδομένων από αρχές, κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμα και από ιδιώτες. Αυτή η μαζική συλλογή στοιχείων και δεδομένων και ε, σε συνδυασμό με κάποιες δηλώσεις ότι είναι για την προστασία συμφερόντων και οικονομικών συμφερόντων αφήνει μεγάλες αμφιβολίες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η στρατηγική παρακολούθηση εξαγωγών όπλων ή τρομοκρατίας, είναι και οικονομικά τα συμφέροντα από πίσω, δηλαδή εμπορική σκοπή. Και εδώ τίθεται το εξή ερώτημα για μένα. Ε, όλα όταν γίνεται επεξεργασία, ανάλυση των στοιχείων και αξιοποίηση. Εκεί υπάρχει έλεγχος και μπορεί το οποιοδήποτε ελεγκτικό όργανο να παρακολουθήσει με ασφάλεια για ποιο σκοπό έχουν συλλεγεί και αξιοποιούν αυτά τα στοιχεία. Και ένα δεύτερο, μιλήσατε πολύ για μηχανισμούς, αρχές και οργανισμούς. Και σε σχέση με την NSA όμως είναι πολλές ιδιωτικές εταιρείες που ενέχονται και στη συλλογή και στην ανάλυση των δεδομένων. Εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος το αργότερο. Αφήστε τις υπηρεσίες. Όταν μπαίνουν ιδιωτικές εταιρείες στη μέση δεν θα πρέπει να ελέγχονται. Um, to begin with, yes. Ε, για να ξεκινήσω, να σε χώρες όπως τις ΗΠΑ ή το Ρωμένο Βασίλειο υπάρχει αυτή η το ηνωμενο βασιλειο υπαρχει αυτη η δυνατοτητα να συγκεντρώνονται δεδομένα και για την οικονομική ευημερία της χώρας. Όπως είπα και στην ομιλία μου, αυτό θα πρέπει να πάψει. Όμω κάποιε εξαιρέσει πρέπει να προβλεφθούν, διότι υπάρχουν και οικονομικά ζητήματα που δίκαιο είναι να αποτελούν αντικείμενο συγκέντρωση στοιχείων. Οι υποψίε οικονομική κατασκοπία εδώ βέβαια είναι άσχημε σε πολλέ περιπτώσει. Έπειτα και για του Γερμανού ή λόγω χάρη για του Σουηδού και του μηχανισμού εποπτεία που διαθέτουν. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να μην είναι τέλειοι, μπορεί να βελτιωθούν, να ενδυναμωθούν με διαφορετικού τρόπου. Όμω αυτοί οι φορεί εποπτεία έχουν πρόσβαση στα γερμανικά ή τα ανάλογα σουηδικά πρότυπα συλλογής. Ε, δηλαδή βλέπουν τι υλικό συγκεντρώνεται και τι όχι. Άρα περισσότερο το πρόβλημα είναι πρόβλημα DNSA. Και σε μικρότερο βαθμό των ίδιων των υπηρεσιών. Ευχαριστούμε. Κοιτάζω αν κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Άγκστρομ, κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι, εντάξει. Εάν ναι, να σας ευχαριστήσω καθηγητά Κάμερον για την σημερινή σας προσέλευση. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για το έργο της Επιτροπής σας και ελπίζουμε να συνεχίσετε στην διπορία. Σα Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσία σας σήμερα. Είναι σημαντικό να μπορούν οι βουλευτές να ακούσουν τα στοιχεία που μας είπατε και μας, αφορά πολύ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό για τους σκοπούς της εποπτείας που συζητούμε σήμερα. Συνάδελφοι, θα αλλάξουμε τώρα ομιλητές. Θα έχουμε τις ομιλίες του κυρίου Λί, του κυρίου Βίλς. Ο κύριος Βίλς συγκεκριμένα μάλλον δυσκολεύτηκε λίγο στο ταξίδι του. Αυτό μου λένε. So Ian Lee is coming up. Οπότε περιμένουμε τον κύριο Λί. Uh, uh, okay. So, hi.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 στο Πανεπιστήμιο του Ντεραμ. Θα μιλήσει εκπροσωπώντα και τον εαυτό του και τον κύριο Βίλ, ο οποίο δυστυχώ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Έχασε το διαβατηριό του, τόσο απλά. Ο Ιαν είναι ειδικό στον τομέα του κοινοβουλευτικού ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών με πολλά άρθρα και μελέτε δημοσιευμένα στο θέμα αυτό και θα μα πει πώ η διεθνή συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών διαφορετικών χωρών ε, εξελίσσεται γοργά χάρη στι τεχνολογικέ ε, εξελίξει επίση και την τεχνολογία για τα δεδομένα. Ε, επίση θα δούμε τι αντίκτυπο υπάρχει στην, εθνικό κοινοβουλευτικό, στην εθνική κοινοβουλευτική εποπτεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχυθεί αυτό το είδο εποπτεία. Έχετε το λόγο κύριε Λίλη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην επιτροπή σα σήμερα. Μου ζητήθηκε από τον κύριο Wills να εκπονήσω εγώ την κοινή μα ομιλία. Και βεβαίω εκ μέρου του συγγνώμη, συγγνώμη που δεν μπορούσε να έρθει. Τελευταία στιγμή αναβολή. Μετά από κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσει για την εποπτεία και την διεθνή και εθνική συνεργασία, στον τομέα τη εποπτεία, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρει τομεί. Θα ήθελα να μιλήσω για τι προκλήσει τη συνεργασία των ε, μυστικών υπηρεσιών σε διεθνέ επίπεδο σε σχέση με του φορεί εποπτεία, τα θετικά βήματα που έχουν κάνει οι φορεί εποπτεία για να ενισχύσουν αυτό το τη συνεργασία και μετά να περάσουν σε κάποιε συστάσει για την εποπτεία σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο. συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών, τα προγράμματα κοινή εποπτεία και η κοινή ανάπτυξή τους, αλλά και ε, οι τεχνολογίες και το πώ κατανέμονται, είναι μέρη και τμήματα της συνεργασίας ε, σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε διεθνές επίπεδο. Όλα αυτά βεβαίω αφορούν άμεσα το θέμα που εξετάζει η Επιτροπή, η ε, δεν θα ασχοληθούμε βεβαίω με τι διάφορε κατηγορίε εδώ ή εικασίε, αλλά θα μιλήσω για το πώ οι φορεί εποπτεία μπορούν να εξετάσουν τα ζητήματα συνεργασία, να τα προωθήσουν. Θα επικεντρωθώ στους μόνιμους φορεί εποπτείας για να δούμε και το ρόλο των δικαστηρίων ή τι γίνεται με επιτόπιες έρευνες στον εσωτερικό έλεγχο. Σημαντικά στοιχεία όλα αυτά. Σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε ενθυμούμενοι ότι η πρόκληση της αντιμετώπισης διακρατικών απειλών από δίκτυα τρομοκρατίας ή την διάδοση των μαζικών όπλων καταστροφής ή του οργανωμένου εγκλήματος, όλα αυτά αναγκάζουν τις μυστικές υπηρεσίες διαφορετικών χωρών να συνεργάζονται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή του η συνεργασία βοηθά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσώπων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία αυτών των χωρών που συνεργάζονται. Ωστόσο, είδαμε από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 το πεδίο και την κλίμακα της συνεργασίας μυστικών υπηρεσιών να εντείνεται και μάλιστα με τρόπο πολλαπλασιαστικό. Η γοργές τεχνολογικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα το να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και δεδομένα γενικότερα, όπως γνωρίζει και μελετά κιόλας το θέμα αυτό η Επιτροπή σας. Στον τομέα της εποπτείας, η διεθνή συνεργασία είναι κάτι που είναι παγιωμένο εδώ και πολύ καιρό. Τα κράτη συνεργάζονται στη συγκέντρωση και την ανάλυση ε, μυστικών πληροφοριών, αλλά και στην ανάπτυξη συστημάτων και υποδομής για αυτούς τους σκοπούς. Το πλέον γνωστό παράδειγμα, που ίσως το ξέρετε όλοι, είναι η συνεργασία ΗΠΑ Βασιλείου Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμαχία που έχει καταρτιστεί από μια σειρά από συμφωνίε τη δεκαετία του 40 και του 50 του περασμένου αιώνα. Προσφατότερα οι μέθοδοι επικοινωνίας και εποπτείας, ε, οι παρακολούθησης έχουν ε, μεταβληθεί δραματικά. Οι βασικοί λόγοι λοιπόν για συνεργασία στον τομέα της εποπτείας έχουν παραμείνει παρόλα αυτά λίγο πολύ αμετάβλητοι. Οι μυστικές υπηρεσίες που έχουν γεωπολιτικά κοινά συμφέροντα συνεργάζονται προκειμένου να αποφεληθούν από την τεχνογνωσία που διαθέτουν τις γεωγραφικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες που μπορεί να ανταλλάξουν. Η εποπτεία, εφόσον βασίζεται στη συνεργασία, δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες για την εποπτεία. Δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την κατανομή εντολών, δηλαδή να είναι κανείς ε, βέβαιος ποια φορέας είναι υπεύθυνο γιατί και βεβαίως δημιουργούνται και κίνδυνοι που ήδη ε, αναφέρθηκαν. Κίνδυνοι που μπορεί τελικά να οδηγήσουν στην παράκαμψη εθνικών ε, προγραμμάτων προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την έγκριση και την ε, οργάνωση της ε, παρακολούθησης ή της εποπτείας. Μπορεί να λαμβάνουν οι μυστικές υπηρεσίες ε, μια σειρά από πληροφορίες που να μην μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις η δομή πρέπει να είναι κοινή, ώστε η ανταλλαγή να γίνεται αυτομάτως οι πληροφορίε μπορεί να παραλαμβάνονται από ξένου συνεργάτε, αλλά θα πρέπει προηγουμένω να έχει υποβληθεί συγκεκριμένο αίτημα. Τώρα, για την εποπτεία, την κοινοβουλευτική εποπτεία εντάχει, μιλήσαμε γι' αυτό. Είπαμε ότι βασίζεται σε κάποιες επιτροπές και τα εξήγησε και ο κύριος Κάμερον, αλλά για τους δικούς μας σκοπούς μπορούμε με αδρό τρόπο να διακρίνουμε τα κοινοβουλευτικά συστήματα εποπτείας και την εποπτεία από ειδικού. Η κοινοβουλευτική εποπτεία κυρίως διεξάγεται από εθνικές κοινοβουλευτικέ επιτροπές, ενώ οι φορείς εμπειρογνωμόνων ή ειδικών από μη ε, βουλευτικούς εκπροσώπους, από ειδικού που σκοπό έχουν αποκλειστικά να εξετάζουν ε, ε, εξονυχιστικά το έργο των μυστικών υπηρεσιών πολλές φορές αυτοί οι ε, φορείς οι ειδικοί μάλιστα ε, αφοσιώνονται περισσότερο και από την άποψη του χρόνου στην ε, σωστό έλεγχο του έργου των μυστικών υπηρεσιών, κυρίως γιατί αυτό είναι το βασικό τους, η βασική τους δουλειά, όχι όπως οι βουλευτές που ίσως για αυτούς να είναι ένα πάρεργο, και έχουν και καλύτερη πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες. Όπως είπα, υπάρχει ποικιλομορφία των ε, προτύπων εποπτείας στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά λίγες είναι οι χώρες που έχουν δώσει σαφή εντολή για τη ρύθμιση των δράσεων και δραστηριοτήτων συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Και μάλιστα σπάνιο είναι να υπάρχει θετική νομοθεσία. Να στραφώ σε κάποιες από τι προκλήσει τώρα τη εποπτεία ε, τη ε, και της συνεργασίας ως προς την εποπτεία. Η βασική δυσκολία είναι ότι εθνική, τα εθνικά συστήματα εποπτείας κυρίως δημιουργήθηκαν προκειμένου να ασχοληθούν με την περίπτωση εγχώριας κατάχρησης ή εσωτερικών παραβιάσεων από τις ε, εθνικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά από την 11η ε, Σεπτεμβρίου και μετά βγήκαμε από την εγχώρια, την εσωτερική αρένα και οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται πλέον σε διεθνές επίπεδο. Να σας πω κάποια από τα βασικά αίτια. Το θέμα που, έχει, που είναι κοινό όλα αυτά είναι η ευκολία πρόσβασης στις ε, ανάλογες πληροφορίες. Όταν η εποπτεία ε, βασίζεται σε πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Ή κάποια ψευδέστηση ότι τα πάντα είναι εντάξει, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όπω είπε ο κ. Κάμερον βεβαίω, εκεί που υπάρχουν δυσκολίε με την πρόσβαση είναι το τι γίνεται με τα τρίτα μέρη. Δεν θα τα εξηγήσω πάλι από την αρχή, αλλά θα μπορούσε κανεί να πει ότι νομικές μνήε για τον κανόνα πρόσβασης τρίτου μέρου η αρχή ελέγχου όπως ονομάζεται, είναι κάτι που συχνά απαντάται στην εθνική νομοθεσία. Αυτό όμω αναστελεί τον τρόπο που οι εθνικοί φορεί εποπτείας μπορούν να διεξάγουν τον έλεγχο των ε, μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Στην πραγματικότητα τι σημαίνουν όλα αυτά. Ότι προτού ο εθνικός φορέας εποπτείας παράσχει πληροφορίες στους επόπτες του, πρέπει να ζητήσει άδεια άδεια από, τους συνεργαζόμενους, από τις συνεργαζόμενες μυστικές υπηρεσίες. Είναι για να το πω αλλιώ. Ε, μια από τις επιπτώσεις είναι να ασκήσουν βέτο οι ξένες μυστικές υπηρεσίες για την εθνική εποπτεία και τις σχετικές δραστηριότητες. Υπάρχουν βεβαίω κάποιε χώρε που αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό, πιστεύοντα ότι δεν θα πρέπει να, παρα, παρεμποδίζει ο κανόνα του τρίτου μέρου ε, και τη αρχή ελέγχου του τρίτου μέρου τη διαδικασία εποπτεία. Είναι τη άποψη ότι οι πληροφορίε που έχουν ε, γίνει κοινέ μεταξύ μυστικών υπηρεσιών έχουν ε, ακριβώ κοινοποιηθεί βάσει αυτών των κανόνων της εποπτείας. Οπότε πληροφορίε που έχουν αποσταλεί δεν θεωρούνται πληροφορίε που ανήκουν στο τρίτο μέρο. Αυτό έχει να κάνει με το πώ αντιλαμβάνονται οι μεν και οι δε τον κανόνα του τρίτου μέρου. Δηλαδή, πληροφορίε που μοιράστηκε κάποιο με μυστική υπηρεσία άλλου κράτου δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη χώρα. Αλλά ο κανόνα του τρίτου μέρου μπορεί να γίνει αντικείμενο κατάχρηση. από τον φορέα, από τη μυστική υπηρεσία μάλλον, προκειμένου να μην υπάρξει πρόσβαση από τον αποπτικό φορέα. Θα μπορούσε μια υπηρεσία να απαντήσει όχι, ε, πολύ απλά, λόγω του φόβου του ελέγχου. Τρίτο μειονέκτημα, η περιορισμός στο τι μπορούν να κάνουν οι εθνικοί φορεί ω προ την εποπτεία και τι δράσει συνεργασία, είναι ότι τι περισσότερε φορέ προσοχή δίνεται στι δικέ του μυστικέ υπηρεσίε. Συμπεριλαμβανομένων των δράσεων των υπηρεσιών αυτών για τις οποίες ενδιαφέρεται και η Επιτροπή σας. Δεν έχουν το δικαίωμα να ερευνήσουν τι δράσει ξένων μυστικών υπηρεσιών οι υποπτικοί φορεί, ακόμη και αν υπάρχει σχέση συνεργασία με, με τις Δεν υπάρχει ούτε εντολή ούτε η νομική εξουσία για να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να αποσπάσουν τι απαραίτητε πληροφορίε από ξένες μυστικέ υπηρεσίες ή ξένου φορεί. Τρίτη δυσκολία είναι το περίπλοκο των προγραμμάτων εποπτείας τα οποία συζητούμε. Κάποια από τα ευρύτερα αυτά συστήματα εποπτείας έχουν τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών με τρόπο αυτοματοποιημένο. Είναι πολύ δύσκολο οι εξωτερικοί επόπτες να τα καταλάβουν όλα αυτά. Ακριβώς το ίδιο και οι επόπτες να τα ρυθμίσουν ή να βρουν νομικές ρήτρες που να έχουν νόημα. Βεβαίω, η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών μεταξύ χωρών είναι αντικείμενο διαφορετικών διτάξεων στι εθνικέ νομοθεσίε. Σε μερικέ χώρε υπάρχει ευρεία ε, αδειοδότηση και είναι πολύ γενικέ οι εντολέ που δίνονται στι μυστικέ υπηρεσίε, το ότι μπορούν να ανταλλάξουν με του εθέρου του. Σε μερικέ περιπτώσει υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει που πρέπει να πληρούνται για να είναι πλήρης η συνεργασία, για κάποιε μορφέ συνεργασία. αλλά πιθανό είναι η παράληψη της αναφοράς της διεθνούς συνεργασίας να μην είναι θέμα ασυνέπειας, είναι απλώς ότι όταν το νομοσχέδιο εγκρίθηκε, όταν πέρασε ο νόμος, να μην υπήρχε πλήρη συνέστηση του ότι ε, διεθνή συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Μπορεί δηλαδή να είναι μια αυλεψία. Να περάσω τώρα στα θετικά βήματα της διεθνούς συνεργασίας. Τι θα μπορούσε να γίνει επιπλέον για την εποπτεία και τη συνεργασία των φορέων εποπτείας μεταξύ τους. Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων είναι ένας χώρος όπου πρέπει να επικεντρωθούμε λόγω των διάφορων ε, ανησυχιών περί ανθρωπινών δικαιωμάτων. Για τον ίδιο λόγο είναι κέρια σημασίας η εποπτεία από το εξωτερικό προς την ανταλλαγή δεδομένων από ε, έναν φορέα με τους συνεργαζόμενους φορείς, αλλά και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται να οριστούν με σαφήνεια. Οι επόπτες θα πρέπει να δουν ζητήματα όπως το εάν η ανταλλαγή δεδομένων εφαρμόζονται, μάλλον συνάδουν με τους ε, ισχύοντες νόμους, το σκοπό για τον οποίο ανταλλάζονται τα δεδομένα, το πώς καλύπτονται οι απαιτήσει περί αναλογικότητας, το αν υπάρχει ε, συγκεκριμένο αρχείο, αν τηρούνται αρχεία για την ανταλλαγή των δεδομένων, εάν υπάρχουν απαγορεύσεις, περιορισμοί και πού έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και αν υπάρχουν απαραίτητες εγγύησεις από τις ξένες συνεργαζόμενες υπηρεσίε. Μια χώρα που έχει αναπτύξει ιδιαίτερα το μοντέλο της για τα θέματα αυτά, που θα ίσως κάτι που θα θέλει να δει η Επιτροπή σας, είναι ο φορέας της Νορβηγίας, η Επιτροπή EOS, η οποία είναι υπεύθυνη για τις νορβηγικές μυστικέ υπηρεσίε. Συχνά πραγματοποιούνται έλεγχοι του πώ ανταλλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα. Αποτιμάται το πού απεστάλησαν τα δεδομένα, εάν η υποκάλυψη των δεδομένων έγινε για νόμιμους σκοπούς, και αν αυτά συνάδουν με τις απαιτήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, πέραν τις ανταλλαγές πληροφοριών που αποστέλλονται εκτός, το ίδιο σημαντική είναι η εποπτεία, και θα έπρεπε να είναι, για την παρακολούθηση του τι γίνεται με τις πληροφορίες που παραλαμβάνονται από τις μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας. Υπό αυτήν την έννοια μπορούν οι υπόπτες να επικεντρωθούν στα αιτήματα για αποστολή πληροφοριών, που έχουν αποστείλει μαλλοντικές τους μυστικές υπηρεσίες σε ξένους εταίρους, για να λάβουν πληροφορίες και ένα σημαντικό θέμα ως προς αυτού του είδους την ε, έρευνα την εποπτεία είναι το κατά πόσο έχει αποσταλεί έτοιμα για πληροφορίες, πληροφορίες που νομίμως έχουν συγκεντρώσει οι ξένες μυστικές υπηρεσίες ή βάση εντάλματος, με ή χωρίς ένταλμα. Οι επόπτες μπορεί επίσης να θέλουν να ελέγξουν κατά πόσον οι παραλαμβανόμενες πληροφορίες εξολογούνται σωστά και κατά πόσον ε, σημαίνονται σωστά, υπάρχει σωστή επισήμανση πρωτού αποθηκευτούν. Το πώς ε, διαχειρίζονται επόπτες τις ε, παραλαμβανόμενες, τις αποστελόμενες πληροφορίες είναι σημαντικό ως προς τις μελέτες αντικτύπου που πραγματοποιούν οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες. Προτού ξεκινήσουν εταιρικέ σχέσεις ή συμφωνίες με άλλες μυστικές υπηρεσίες. Ένα καλό παράδειγμα για αυτά στην πράξη είναι η διεξοδική μελέτη που γίνεται σχετικά από τον φορέα Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, το CTIVD, το οποίο από το 2009 καθιέρωσε τις ε, θεματικές εκθέσεις για την επίβλεψη της ε, διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών. Επιτρέψτε μου τώρα να, στραφώ, να περάσω σε κάποιες συστάσεις και για το εθνικό επίπεδο και ίσως λίγο συντομότερα για το ευρωπαϊκό. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουν οι εθνικοί φορείς εποπτείας. Αυτοί είναι οι κατεξοχήν πρωταγωνιστές στην ε, παρακολούθηση των διαδικασιών συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και για να δουν κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν με το κράτο δικαίου, την νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εθνικοί υπεύθυνοι φορείς έχουν και την εντολή και την καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και μπορούν να υπερβούν τις δυσκολίε. Το, η λογοδοσία λοιπόν εξασφαλίζεται ενισχύοντας το ρόλο των εθνικών φορέων που κοιτάνε τις διαδικασίες συνεργασίας. Το βάρος της ευθύνης λοιπόν το έχουν οι εθνικοί νομοθέτες από αυτή τη λογική. Οι υπάρχοντες φορείς εφόσον λειτουργούν σωστά στον τομέα αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν. Εκεί που χώρες, υπάρχουν χώρες χωρίς ε, την ε, εποπτεία από ειδικού για τις μυστικές τους υπηρεσίε. Τι χρειάζεται. Ε, είναι προφανές ότι οι κοινοβουλευτικοί φορείς δεν αρκούν. Καλό λοιπόν θα ήταν να διορθωθεί αυτό. Σε χώρες όπως το Βέλγιο, τις κατοχώρες τη Σουηδία. Να χρησιμοποιηθούν αυτές ως παράδειγμα και να υπάρχει ένας φορέας εμπειρογνωμόνων που να συμπληρώνει το κοινοβουλευτικό έργο εποπτείας. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Πώς αποτιμάται η αποτελεσματικότητα των ε, διαδικασιών εποπτείας. Αυτό νομίζω δεν θα το ε, απαντήσω εδώ. Να στραφώ στο τι μπορεί να κάνει η νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο και τι όχι. Ένα στοιχείο θα ήταν να υπάρχει κάποια μνήα για την εποπτεία και τη διεθνή συνεργασία στις εγχώρες νομοθεσίες. Εκεί που απαντάτε ε, εντάξει, αλλά κάποιες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το έχουν καλύψει το θέμα αυτό, κάποιες άλλες όχι. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι η εθνική νομοθεσία έχει και τα ωριά της. Δεν μπορεί να ρυθμίσει το τι θα κάνουν οι ξένοι, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται μια χώρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ρυθμίσουμε τουλάχιστον την διαδικασία, τη μέθοδο με την οποία συνάπτεται κάποια μορφή συνεργασίας με ξένες μυστικές υπηρεσίες, ώστε τουλάχιστον αυτό να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσει του δικαίου και τον σεβασμό τι απαιτήσει του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα βήμα πρόοδου θα ήταν να δημιουργηθεί ένα ένας κατάλογος από κριτήρια για αυτές τις συμφωνίες συνεργασία και τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται. Μια σειρά από φορείς έχουν συστήσει αυστηρότατα νομοθετικά πρότυπα στον τομέα αυτό, στον χώρο αυτό, η Διεθνής Επιτροπή Νομικών Ειδικών και ε, ένα σώμα νομικών εμπειρογνωμόνων. Το πρώτο είναι αυτό το 2009 μέσω του ε, ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ, που και αυτός έκανε ανάλογες συστάσεις. Επίσης, ε, υπάρχουν άλλες αναφορές της καταληκτήριες παρατηρήσεις μου, αλλά δεν θα διμείνω, για τις προτάσεις της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά. Όπως είπα προηγουμένως, το δεύτερο βήμα πρόοδου θα ήταν να αντισταθούμε στην ιδέα ότι ο κανόνας του τρίτου μέρους θα έπρεπε να παρεμποδίζει τους επόπτες. Δηλαδή, εάν τέτοιοι κανόνες υιοθετηθούν, οι φορείς εποπτείας δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως τρίτα μέρη ευθύς εξ αρχής. Οπότε να μην χρειάζεται καν άδεια προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συνεργαζόμενων ε, φορέων. Εάν αυτό ήταν το σημείο αφετηρίας, θα ενισχυόταν και η εποπτεία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλο, επειδή οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται ούτως ή άλλως με ομόλογες μυστικές υπηρεσίες σε άλλε χώρε, γιατί να μην μπορούν και οι φορεί να κάνουν το ίδιο, οι φορεί εποπτείας. Τι εννοώ, δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχουν κοινέ έρευνε. Ναι. Ίσως αυτό υπερβαίνει κάπως τα όρια των όσων έχουμε σκεφτεί ως τώρα ή των όσων προβλέπουν οι νομοθεσίες, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινά συστήματα, όπου οι επόπτες σε μια χώρα που θέλουν να περάσουν σε μια κοινή έρευνα, η κοινή παρακολούθηση, να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο φορέα της ε, εν λόγω χώρας που τους ενδιαφέρει και να ζητήσουν συμπληρωματικές εκθέσεις, να αποκάλυψει στοιχείων. Αυτά είναι βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Τώρα τι μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ να υποστηρίξω την ε, ιδέα που ανέφερε ο κ. Κάμερον ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη σύγκληση, στην συνέχιση μάλλον τη ε, σύγκληση συναντήσεων ε, των εθνικών εποπτικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι μπορούν να ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, να παίξει έναν επιπλέον ρόλο στην προώθηση των ελάχιστων προδιαγραφών για τις ε, καλές πρακτικές, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει ο ειδικό εισηγητή ε, του ΟΗΕ και η Επιτροπή τη Βενετία. Θα δίσταζα βεβαίω να αποδεχτώ με άνεση την ιδέα ότι θα πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα. Να εξελιχθεί δηλαδή το σύστημα των κοινών συναντήσεων σε ένα φόρουμ για την πραγματική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μου φαίνεται ότι θα παρουσίαζει αρκετέ νομικέ δυσκολίε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Εμεί σα ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά μου. Είναι βέβαια 4 η ώρα, 5η απόγευμα. Αναρωτιέμαι ποιο παρακολουθεί τους κανόνες με τους οποίους δίνουμε το λόγο στη συζήτηση. Ο Γιάνν Άλμπρεχτ πρώτος. Ευχαριστώ Κλάβδιε. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την παρουσία σας. για τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε για να βελτιώσουμε τη αντιμετώπιση της παρακολούθησης των πολιτών. Λέγεται ότι συνεργάζονται όσοι παρακολουθούν, αλλά ότι επίσης η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών σημαίνει και ανταλλαγή πληροφοριών και ότι αυτό είναι από τους απαράβατους κανόνες. Επομένως, εδώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την δομή που έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη μας λένε συνεργαζόμαστε για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών ως προς την εθνική ασφάλεια αλλά στέλνουμε και επιστολά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου δεν σχολιάζουμε τα εσωτερικά μας και δεν θα έρθουμε να μαρτυρήσουμε ούτε θα δεχτούμε κοινά πρότυπα ή κανόνες Αυτά δεν συνδυάζονται μεταξύ τους και επίσης από την άποψη που δουλεύουμε εμείς εδώ τα κράτη-μέλη δεν σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ μυστικών υπηρεσιών αλλά θεωρούν ότι δεν μειώνονται έτσι οι εθνικές τους κυριαρχίες. Τι λέει. Το δεύτερο ερώτημα. Όταν γίνονται αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών, πώς μπορεί να το ελέγξει αυτό το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού ούτε καν τα εθνικά δεν μπορούν. Uh, is for the other one because... Ξέρουμε ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας και το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ελέγξει παρά μόνο τη δική του μυστική υπηρεσία, όχι του άλλου κράτους. Είναι λοιπόν, γίνεται λοιπόν φανερό ότι με το υπάρχον σύστημα αν δεν αλλάξουν οι κανόνες, αν δεν έχουμε καινούργιες ιδέες για το πώς να γίνει αυτή η επιτήρηση, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ. τονίσατε δύο βασικές ε, δυσκολίες. Εγώ δεν είμαι ενωσιακός δικηγόρος. Ε, απλώς αναγνωρίζω την πραγματικό, τις πραγματικότητες. Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι ισχύει ήδη εδώ μέσα. Το προφανές είναι ότι πολλές από αυτές τις διευθετήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι διμερείς, πολύ σπανιότερα πολυμερείς, αλλά όχι συλλογικές. το δεύτερο που είπατε, μάλιστα τα εθνικά κοινοβούλια δεν βλέπουν παρά μόνο αυτά που κάνουν οι δικές τους υπηρεσίες το καθένα. Και νομίζω ότι τα κοινοβούλια δεν είναι το καλύτερο μέσον τα καλύτερα πρότυπα είναι η ρεαλιστική εξέταση από εμπειρογνώμονες που έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση στα στοιχεία και μπορούν να τα ελέγξουν. ενώ οι κοινοβουλευτικές επιτροπές είτε απαιτούν έγγραφα και μαρτυρίες από υπαλλήλους είτε όχι, μπορεί να μην είναι σε θέση τόσο να το πράξουν. Στο Βέλγιο ξέρω ότι χρησιμοποιούνται πολλοί εμπειρογνώμονες και στην Νορβηγία. Πολύ παραπάνω από ό,τι σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κορνιλία Χέρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Τρία πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Πρώτον, όλα αυτά που μας είπατε, αλλά και οι προλαλήσαντες εμπειρογνώμονες αναφέρθηκαν σε αυτά, έχω την αίσθηση, πώς να το πω, ότι είναι λίγο ο λαγός με τη χελώνα, για να πω και το μύθο που γνωρίζετε. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι είμαστε μια χελώνα, ε, τα αποεπτικά, όργανα και τρέχουμε και η λαγή που είναι οι μυστικές υπηρεσίες με όλη την τεχνολογία που έχουν και τη δυνατότητα μας έχουν αφήσει πίσω. Θα πρέπει να γνωρίζει ο επόπτης ε, και τα τεχνικά πραγματικά για να μπορεί να ελέγχει. Για μένα είναι γενικότερο αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν πρόκειται οι μυστικές υπηρεσίες να θελήσουν να υποβληθούν σε έλεγχο, το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει αυτό το έλλειμμα της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων. Είπατε κάτι ε, ε, που υποστηρίζω και εγώ, ότι χρειάζονται ε, και σώματα εμπειρογνωμόνων συμπληρωματικά προς το Κοινοβούλιο, συμφωνώ. Αλλά ποια θα είναι η σύνθεση αυτών, εσείς πώς το βλέπετε, οι επόπτες προσωπικών δεδομένων, οι εθνικοί, οπωσδήποτε, αλλά εκτός από αυτούς, ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν εκεί και πώς θα έχει συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, ε, σήμερα το πρωί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ούτε να φλιαρίσω, αλλά συζητήσαμε με τον Ίνθισεν. θα μπορούσατε κάπως να αξιολογήσετε το δικό τους ε, ρόλο. Ε, τους βλέπετε να συμμετέχουν κάπως εκεί στον έλεγχο. Ε, πώς το φαντάζεστε. Yes, I, your remarks about the uh, Χαίρομαι για τα σχόλια σας, σας προς την περιπλοκότητα ε, αυτών που καλούμαστε να εποπτεύσουμε στην παρακολούθηση. Θα μπορούσαν οι οργανισμοί ε, εποπτείας να χρησιμοποιήσουν και εξωτερική πραγματογνωμοσύνη για αυτά τα τεχνικά, για ορισμένα, εν πάση περιπτώσει. Ε, και οι ε, καταγγέλλοντες, οι λεγόμενοι whistleblowers, θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για τέτοιου είδους έρευνες. Ως πληροφοριοδότες δηλαδή. Τώρα για τα σώματα εμπειρογνωμόνων και πώς έρχονται αυτά να συμπληρώσουν το κοινοβούλιο. Εμείς τι θέλουμε. Να είναι πολιτικά όργανα που να έχουν δηλαδή επαρκή ε, ε, νομική και τεχνική δυνατότητα ή στελέχωση, εν που να μπορεί να τους πλησιώνει και να τους βοηθάει για τέτοιου είδους ελεγκτικό έργο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι, όχι μια επιτροπή σοφών με ε, βετεράνους, ηγέτες, άνδρες ή γυναίκες, αρχηγούς κρατών. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται και πιο ειδική γνώση για να γίνεται ε, ουσιαστικός έλεγχος σε αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά την Ίντσεν, εγώ δεν είμαι ειδικό στο ευρωπαϊκό δίκαιο και το λέω με επιφύλαξη, θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για να έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο ε, εάν είναι εντός τη της εντολής που έχει λάβει και των νομικών ε, εξουσιών. Εκεί μπορεί να υπάρχει κάποια δυσκολία. Ευχαριστώ. Η Μπριγκίτ Σίπελ. Θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω κάτι στα γερμανικά. Δεν είμαι βέβαια ότι σας κατάλαβα καλά προηγουμένως αυτό που μας είπατε. Εγώ κατάλαβα ότι ο νομοθέτης καμιά φορά δεν έχει ιδέα για τις ε, διαστάσεις του φαινομένου, σε ποιο βαθμό συλλέγουν πληροφορίες οι μυστικές υπηρεσίες. Και διαρωτώ με, αν δεν έχει ιδέα ο νομοθέτης, δεν μπορεί και να ελέγξει με σωστό τρόπο. Γιατί δεν έχει ιδέα λοιπόν ο νομοθέτης, γιατί δεν γνωρίζει τι δυνατότητες υπάρχουν και τι δραστηριότητες διεξάγονται και πώς θα κληθεί να τα ελέγξει όλα αυτά αν δεν έχει ιδέα. Αλήθεια είναι αυτό ότι πάντα θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Και η δεύτερη ερώτηση, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να την απαντήσετε εσείς. Εδώ μιλούμε για την εργασία των μυστικών υπηρεσιών που κατά κανόνα εκτός ε, ορίων της επικράτειας της χώρας τους ε, μαζεύουν στοιχεία, αλλά τους ίδιους δεν θέλουν να τους παρακολουθούν. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για ποιο, ποιος είναι αρμόδιος για την αντικατασκοπία. Υπάρχουν ενιαίες ρυθμίσεις, υπάρχουν ε, ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων μυστικών υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών, δηλαδή εννοώ την κατασκοπία και την αντικατασκοπία. Και ένα πολιτικό ερώτημα. Πάντα εκπλήσωμαι όταν λένε διάφοροι υπουργοί ότι σιγά την είδηση. Εγώ πάντα θεωρώ ότι μου παρακολουθούν το τηλέφωνο. Και διερωτώ με, ακριβώς για υπουργούς, μα υπουργοί κανονικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εμπιστευτικών συνομιλιών με κάποιους άλλους και απορρίτων. Ελπίζω να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Χωρίς να τους παρακολουθεί κανείς, χωρίς να υποκλέπτει τις συνομιλίες ε, ή να υπάρχουν συνακροάσει. Και πώς μπορείς να κάνεις τέτοια εμπιστευτικά τηλεφωνήματα όταν ξέρεις ότι σε παρακολουθούν και από πάνω. Δεν ξέρω. Αυτά πώς συνδυάζονται. On the Για το θέμα της εμβέλειας και των όσων γίνονται και πώς μπορούμε να καλύψουμε, θα μπορούσα να πω τα εξή δύο. Πρώτον, σε κάποιες χώρες η δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει νομοθεσία, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες χώρες ισχύει έτσι. Ε, Επίτηδες οι νόμοι είναι ε, θολοί και συγκεχημένοι. Mm-hmm. Έχουν συνταχθεί έτσι για να μην καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται και τι τρέχει και τι επιτρέπεται. Αν κοιτάξτε ε, το 2000 την νομοθεσία μας, ας πούμε, το νόμο ε, για τις αρμοδιότητες. Πρέπει να παρακολουθήσει κανείς να διαβάσει τους ορισμούς πολύ προσεκτικά για να καταλάβουμε τι γίνεται με την παρακολούθηση και τι ισχύει και τι ε, επιτρέπεται. Και γι' αυτό πραγματικά εκπλήσωμαι αν ήξεραν ε, οι νομοθέτες τι ψήφιζαν όταν ψήφιζαν τέτοια πράγματα σε μερικές χώρες. Γιατί είναι πραγματικά σκοτάδι αυτό που επικρατεί εκεί. Η εποπτεία που λειτουργεί σωστά όταν υπάρχει εμπιστοσύνη με τις υπηρεσίες. Και έχουν ανταλλαγές προφοριών και δεν τηρούνται μυστικά αυτά τα στοιχεία ε, προς τους επόπτες. Τώρα δεν... Ξέρω, από χώρα σε χώρα διαφέρουν τα συστήματα και δεν μπορούν να δημοσιεύονται και πάρα πολλά πράγματα με τον τρόπο αυτό. Υπάρχουν εμπιστευτικέ ε, πληροφορίε. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για να μην συλλέγονται στοιχεία, είναι πολύ λίγοι νόμοι αυτοί. κανονικά ε, πρόκειται για περιορισμούς ε, στη συλλογή στοιχείων για τους πολίτες μιας χώρας. Και στη Γερμανία νομίζω και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας δεν παρακολουθούν τους ίδιους πολίτες της χώρας, υποτίθεται. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες. Αυτή είναι η πρώτη μορφή περιορισμού που γνωρίζω εγώ, εν πάση περιπτώσει, για τις εμπιστευτικές συζητήσεις μεταξύ πολιτικών πρέπει να σας πω. Εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο από τη μαζική παρακολούθηση των πολιτών παρά των πολιτικών, για να είμαι ειλικρινής. Mm. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Ε, ορισμένες χώρες, τουλάχιστον επίσημα, ε, έχουν ε, προστασία. Ας πούμε στη Βρετανία υπάρχει ένα αντίστοιχο δόγμα και οι Βρετανοί βουλευτές δεν παρακολουθούνται. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, καταλαβαίνετε, που ξεπερνάει τον νόμο. Δεν ξέρω αν έχετε συμπροματικές ερωτήσεις ή λοιπές ή άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν θέλουν. Εντάξει, σε λίγο είπαμε ότι θα μας πείτε τη μαρτυρία σας λοιπόν. Μπορώ να θέσω ένα ερώτημα. Όχι. Ακόμα είναι μόνο για βουλευτάς. Εσείς σε λίγο. Έτσι γίνονται οι ακροάσεις. Τι να κάνουμε. Άννα Γκόμες, ήθελες να θέσεις ερώτημα. Ναι. Κατανοώ την προσέγγιση σας ότι χρειάζεται ειδικευμένο σώμα για να τα δει όλα αυτά πιο αποτελεσματικά στην εποπτεία, δηλαδή την επιτήρηση των υπηρεσιών. Αλλά να δούμε τι έγινε με την προστασία των δεδομένων σε χώρες όπως τη δική μου την Πορτογαλία όπου υπάρχει μια Εθνική Επιτροπή για αυτό το θέμα άκουσε εμπειρογνώμονες άλλους που όρισε το Κοινοβούλιο νομομαθείς και πολλές φορές αντιμετώπισαν καταστάσεις που τις θεώρησαν αντίθετες με την νομοθεσία μας και διαμαρτυρήθηκαν και δεν έγινε τίποτα. Χρησιμοποίησαν τους διάβολους που προβλεπόταν και δεν έγινε τίποτα. Μόνο όταν ατομικά ορισμένα από αυτά τα μέλη ήρθαν σε εμά, στους ευρωβουλευτάς, μόνο τότε βγήκε το θέμα. Και για μας ήταν πολύ δύσκολο. Εμείς δεν είμαστε τμήμα της διαδικασίας αυτής. Επομένως, κερδίζουμε τίποτα άμα δεν γίνονται αυτές οι έρευνες από το Κοινοβούλιο ενώ έχουν την απαραίτητη πολιτική ευθύνη. Με τη βοήθεια βέβαια εμπειροχνομόνων. Εγώ δεν είπα να υποκαταστήσουν οι εμπειρογνώμονες τα δημοκρατικά όργανα και την λογοδοσία αλλά είπα να συνδέονται οι εμπειρογνώμονες με τα όργανα. Δεν έλεγα ή το ένα ή το άλλο. Άλλες χώρες όμως που έχουν μόνο κοινοβουλευτικά όργανα δεν, δεν Μάλιστα κύριε καθηγητά. Προηγουμένως που δεν σας έδωσα το λόγο δεν ήταν από αγένεια, ήταν γιατί οι ευρωβουλευτές είναι παντού εδώ μέσα και έπρεπε να διασφαλίσω ότι θα ρωτήσουν πρώτα όλοι οι ευρωβουλευτές αυτά που ήθελαν γι' αυτό, να, γιατί έτσι το κάνουμε. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Α, σας απάντησε ο άλλος, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά η έλλειψη νομικού πλαισίου είναι κάτι που καθιστά ακόμα πιο πολύτιμη τη συμβολή σας για μας και σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας παρουσίαση. Ευχαριστώ. running ahead of time. Λοιπόν, είμαστε νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρόνο. Ε, έχουμε δύο μάρτυρες τώρα για την επόμενη ε, ενότητα, ο κύριος Μπίκφορτ και ο κύριος Χωσέιν. Ε, ε, είναι το θέμα που αφορά την κατάσταση στον Ηνωμένο Βασίλειο και τους παρακαλώ να έλθουν εδώ στο βήμα. Colleagues, if you want to take your uh, places, we can get started. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να καθίσετε συνάδελφοι για να αρχίσουμε όχι Λοιπόν, αρχίζουμε. Ε, την επόμενη ενότητα που είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και επίκαιρη. Νομίζω για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο η Βουλή των Κοινοτήτων στην αντίστοιχη επιτροπή τη που μιλάει για κοινοβουλευτική εποπτεία, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, θα ακούσει τους επικεφαλείς ε, του MI5, MI6 και GSHQ μαζί όλους αυτούς την ίδια μέρα. Ενδιαφέρον έω σύμπτωση ε, για να δούμε πόσο επίκαιρη είναι αυτή η υπόθεση και πολύ ενδιαφέρον έτσι, που συνέπεσε αυτή η μέρα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο να ακούσουμε τις μαρτυρίες, να αναλύσουμε ε, τι συμβαίνει και καλωσορίζουμε τον κύριο David Beckford που είναι ο πρώην νομικός διευθυντής ε, των Υπηρεσιών Ασφαλείας και Πληροφοριών MI5 και MI6 και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Γκάς Χωσέιν που είναι εκτελεστικός διευθυντής της ε, Privacy International, της Διεθνούς Ιδιωτικής Ζωής. Ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπίκφορτ λοιπόν Are you good, David? Are you going to make anything available to members or present by way of presentation, or are you just yes, I have. Έχετε και παρουσίαση PowerPoint. Έχω, αλλά νομίζω ότι έχει διανεμηθεί ήδη ανέμετα αυτή τη στιγμή. Να σας δώσω τότε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Do that. Yeah, thank you very much for asking me to... Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι η δημόσια γίνεται ακρόαση στην αντίστοιχη Επιτροπή της Βολής των Κοινοτήτων, των Διευθυντών των Μυστικών Υπηρεσιών. Το ζητώ εδώ και χρόνια στην Αγγλία αυτό, ε, από τότε που άρχισε η νομοθεσία να ισχύει, οπότε είναι πολύ καλή ημέρα πραγματικά. Και ακόμα καλύτερο είναι που βρίσκομαι εδώ εγώ. Υπάρχει δημόσια δυσταρέσκεια ε, για τις διοκτικές αρχές και τις μεγάλες εξουσίες τους. Πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση πραγματικότητα αυτό, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ε, μία πραγματικότητα είναι ότι οι εξουσίες αυτές ρυθμίζονται δια νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην αντίστοιχο νόμο του 2000, που έχει και κώδικα δεοντολογίας και ε, χρειάζεται ε, δικαστική άδεια για να γίνονται αυτές οι δράσεις. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, θεώρησε ότι οι διατάξεις και οι πρόνοιες ε, αυτού του νόμου στην υπόθεση Κέννιντι κατά Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούσε κατάχρηση εξουσίας και έγιναν παράνομες υποκλοπές και εδώ απαντώ στον καθηγητή Λί που μιλεί για την ε, περιπλοκή των νόμων και της νομοθεσίας. Μα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υπόθεση Κέννιντι ε, έχει να κάνει και με την υπόθεση κλάς κατά της Γερμανίας ε, του 1978 που επίσης θεωρήθηκε η βάση για δράση των μυστικών υπηρεσιών. Και η εποπτεία ε, πραγματικά ασκήθηκε εκεί με τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η δυσαρέσκεια λοιπόν του κόσμου βασίζεται στην αίσθηση που έχει. Γιατί δεν καταλαβαίνει ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, υπάρχει ισορροπία ανάμεσα ε, στην ιδιωτική ζωή και την κρατική ασφάλεια. Άλλο είναι το αστυνομικό κράτος και άλλο είναι η παρακολούθηση ε, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι δημοκρατικοί θεσμοί. Σήμερα όλο και περισσότερο ε, υπάρχει παρακολούθηση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Και εφόσον ε, επιτρέπουν οι υπουργοί τις υποκλοπές, τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, τις επικοινωνίες λοιπά, Ε, ο κόσμος αμφιβάλλει αν ένα τέτοιο καθεστώς μπορεί να γίνει ανεκτός σε συνθήκες δημοκρατίας. Η πρόταση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ήρθε να περιπλέξει τα πράγματα με μια ανακοίνωσή της, data poll, ε, για ε, την επεξεργασία και συγκέντρωση, των data mining διαφόρων στοιχείων. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν εμπίπτει ακριβώς στις μυστικές υπηρεσίες. Έχει να κάνει με τις διοκτικές αρχές, τα τελωνία, τις υπηρεσίες μετανάστευσης και άλλες. Και η παρακολούθηση ε, πολλές φορές γίνεται ε, χωρίς δικαστική άδεια. Ε, όλοι αυτοί οι οργανισμοί υφίστανται πίεση ε, για την ασφάλεια του κοινού, του λαού και οι ίδιοι υπουργοί πιέζονται. Λοιπόν, με όλη αυτή την πίεση οι υπουργοί όχι απλώς αποφασίζουν την εκτεταμένη παρακολούθηση αλλά αποφασίζουν και την καθημερινή διεισδυτική παρακολούθηση κάθε στόχου. Και περιορίζεται σε αυτό το στόχο. Ε, ε, μυστική παρακολούθηση ε, παρακολουθεί για λόγους ε, εγκλήματος και τρομοκρατίας αλλά συλλέγονται και άλλες πληροφορίες με άλλο τρόπο είναι πάρα πολύ μυστικές, πάρα πολύ ευαίσθητες και τίστε και το δίλημα ποιος μπορεί να γνωρίζει αυτά τα πράγματα και να τα μαθαίνει όλη αυτή η πίεση λοιπόν ε, μπαίνει σε μια ζυγαριά ανάγκης και αναλογικότητας όταν ζητούν την άδεια υπηρεσίας και όταν σκέφτονται να τη δίδουν οι ε, ε, υπουργοί. Στην υπόθεση Κλάς το 1978 δεν υπήρξε πολύ μεγάλη παρακολούθηση, ενώ στην υπόθεση Κένετι είχαμε τηλεφωνικές υποκλοπές ε, από ένα, ένα πρόσωπο που είχε καταδικαστεί για φόνο. Σήμερα βέβαια δεν ισχύουν αυτά τα επιχειρήματα. Όταν υπάρχει τέτοια ευρεία παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες ε, και profiling και data mining, αυτό γίνεται οριζόντια και σε πολύ ε, μεγαλύτερη εμβέλεια που υπερβαίνει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. The court the class decision... Σύμφωνα με την υπόθεση κλάς λοιπόν το δικαστήριο απεφάνθη όταν είναι τόσο εύκολη η κατάχρηση σε μεμονωμένες περιπτώσεις και μπορούν να έχουν τέτοιες επιπτώσεις αρνητικές για την ε, δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει εποπτικός έλεγχος από ένα δικαστή. Το δικαστήριο είπε ιδιαίτερα ότι μεταξύ άλλων κράτος δικαίου σημαίνει ότι όταν η εκτελεστική αρχή μπαίνει σε δικαιώματα ατόμων θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος επαρχικής από τη δικαιοσύνη. Σε τελική ανάλυση ο δικαστικό έλεγχος είναι το καλύτερο εχέγγυο για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη σωστή διαδικασία. Κατά την άποψή μου, και το έχω πει επανειλημμένα αυτό, η ε, εκτεταμένη παρακολούθηση που γίνεται σήμερα και η άδεια που ζητείται. Ιδιαίτερα αν βάλουμε και πάλι στη ζυγαριά την ανάγκη με την ε, αναλογικότητα, μας δείχνει ότι η αρχή της υπόθεσης κλάς για δικαστική άδεια πρέπει να βρει εδώ η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία αν θέλετε, πρέπει να βγει από την εξίσωση και να μπαίνει ε, στα χέρια της δικαιοσύνης και μόνο η διαδικασία έγκρισης. Δηλαδή, η μυστική υπηρεσία θα πρέπει να ζητεί ε, την άδεια από τις δικαστικές αρχές χωρίς να περνάει από την κυβέρνηση για να παγιδεύει τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες και λοιπά. Και για τους πληροφοριοδότες. Αυτή η διαδικασία μειώνει λοιπόν την αίσθηση της διαπλοκής ε, ε, εξαιρεί την κυβέρνηση και δεν υπάρχει χώρος για κατηγορίες εμπλοκής του κράτους ε, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει λοιπόν ανεξάρτητη εποπτεία και το ίδιο το κοινοβούλιο τους εποπτεύει και όπως βλέπετε σήμερα ε, βλέπουμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό. Αλλά και αυτή η εποπτεία, αλλά και ο έλεγχος από ε, το ε, αρμόδιο δικαστήριο γίνεται εκ των υστέρων. Και κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις δικαστικές αρχές. Επίσης, Ε, και στις Ηνωμένε Πολιτείε δίνεται δικαστικός έλεγχος και έγκριση από δικαστές. Ο πρόεδρος Μπούς όμως ε, στον πόλεμο κατά της ε, τρομοκρατίας παρέκαμψε την, τον νόμο Φάι και κατήργησε ουσιαστικά την κανονική λειτουργία που είχε στο παρελθόν. Αν δίνεται όμως δικαστική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο για παρακολούθηση τηλεφώνων και ε, ηλεκτρονικών μέσων, ε, ε ήταν ε, πολύ άστοχο στο γαλλικό σύστημα ο ανακριτής ε, εποπτεύει τις ε, καλυμμένες ε, και μυστικές δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών, τη μυστική παρακολούθηση και η απόφαση 2005 κάθετος 532 της 19ης Ιανουαρίου 2006 είναι κάτι που μας βοηθάει να καταλάβουμε την κατάσταση οι πιέσεις που υφίστανται οι υπουργοί δεν υπάρχουν στην περίπτωση των δικαστών, οι οποίοι επαγρυπνούν να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αναλογικότητας ε, και ιδιωτικής ζωής και προστασίας του κοινού. Επιπλέον ο ανακριτής εποπτεύει την όλη διαδικασία και ε, παίρνει αποφάσεις σε μεταλόγου γνώσεως και πλήρη εικόνα της καταστάσεως. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία και Πραγματικά είναι ενθαρρυντικό να το βλέπει κανείς. Άλλο σημαντικό θετικό του δικαστικού συστήματος είναι ότι σε αντίθεση ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, υπάρχει παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έτσι ε, μειώνονται οι πιθανότητες να γίνουν λάθη και σε συνέχεια παρατράγουδα κατά τη διαδικασία και τις δίκες και αυτό βοηθάει και τις μυστικές υπηρεσίες και τις διοκτικές αρχές. Το σύστημα αυτό του δικαστή που παρακολουθεί την όλη διαδικασία είναι εγγύηση για ανεξάρτητη, μη πολιτική ε, και ε, ψύχρεμη και αντικειμενική εποπτεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε απευθείας στον κύριο Γκάς που είναι ο ε, Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικός Διευθυντής του Πορεία <clears throat> για την ε, εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων. Και έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. <coughs> Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Ναι με τέτοιους ε, μεγάλους ρήτορες που είχαμε απόψε το σήμερα το απόγευμα μαζί μας με τόσες γνώσεις. Να αναφέρω και εγώ τη σημασία της παρουσίασης του κυρίου Πίκφορντ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνουμε μάχη εδώ και 17 χρόνια να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το θέμα της έγκρισης από τους πολιτικούς. Υπάρχει τρομερή αντίσταση στην αλλαγή και την έγκριση της δικαστικής, μάλλον την ε, ανάγκη, την πρόβλεψη απέτησης για δικαστική άδεια. Η, το τέλος της ομιλίας του κ. Μπίκφορτ διεύρυνε κάπως το πεδίο της συζήτησης. Όμως, εγώ από την σκοπιά της εποπτείας θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία, διότι εάν μιλάμε για μόνιμη εποπτεία, δεν θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε σωστά στα όρια του ζητήματο, διότι το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι θέμα εποπτεία, είναι θέμα δικαίου. Έχω λοιπόν τρία σημεία τα οποία θέλω να αναπτύξω. Το πρώτο, πρώτα απ' όλα α θυμηθούμε. Α θυμηθούμε γιατί, προ... για τι είδου προγράμματα συζητούμε. Το πρωί ακούσατε για τα προγράμματα μαζική παρακολούθηση το Τέμπορα, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα με υποθαλάσσια καλώδια που παρακολουθούνται, που μπορεί να υπάρχουν παντού στον κόσμο από θαλάσσια καλώδια και την αποθήκευση την αντιληπτικά μόλι την περασμένη εβδομάδα που η GCHQ ασχολήθηκε με ένα πρόγραμμα μαζική συγκέντρωση δεδομένων από το Google και το Yahoo και τα κέντρα δεδομένων τους. Αντλούσε όσα δεδομένα μπορούσε με επίθεση ουσιαστικά, με ομή επίθεση, α το πούμε έτσι. Επίθεση στα καλώδια που ανήκαν σε αυτέ τι εταιρείε. Αυτό είναι το πρώτο είδος ε, παρέμβασης. Έπειτα υπάρχει η εκμετάλλευση μηχανών ε, εργαλείων και δικτύων. Αυτό περισσότερο μοιάζει με επίθεση παρά με νόμιμη πρόσβαση. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα να στραφεί ένα μηχάνημα εναντίον του χρήστη. Ή ένα ολόκληρο δίκτυο εναντίον του χρήστη. Το ακούσατε από προηγούμενους ομιλητές. Το τρίτο είδος προγράμματος είναι η εκμετάλλευση των πρωτοκόλων ασφαλείας και των προτύπων ασφαλείας. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό κατά την άποψή μου. Διότι εδώ αυτό μπορεί να συνεχιστεί ακόμη για να αλλάξουμε τους νόμους. Δηλαδή, η NSA και η GCHQ έχει, έχουν παραβιάσει τα πρωτόκολλα. Με χρηματοδότηση, με συγκεκαλυμμένη ε, επιρροή στο τι σχεδιασμό προϊόντων κάνουν οι εταιρείε. Αυτά Πόρο απέχουν από την νομική εποπτεία ή την ε, παροχή άδεια ή την ε, γνώση υπουργού ή δικαστηρίου. Μιλάμε για πραγματικό σαμποτάζ των πρωτοκόλων ε, ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες εταιρείε παγκοσμίω. Από κοινού τα προγράμματα αυτά ουσιαστικά πλήττουν τα θεμέλια και τα συστήματα στα οποία βασιζόμαστε για τον προσωπικό, τον επαγγελματικό, τον εμπορικό μας βίο και την ευημερία μας. Γι' αυτό μόλις χθε το Τέμπορα επιτέθηκε ακριβώ στα προγράμματα αυτά, αποκαλώντας τα ε, και ανόητα και αποτρόπαια. Ας ε, τώρα στο International, επικεντρωνόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια από τις πρώτες μας δράσεις ήταν να προσφύγουμε κατά της κυβέρνησης για τη συνεργασία της στο πρόγραμμα PRISM, αλλά και στο Tempora. Ρωτήσαμε ένα απλό, θέσαμε ένα απλό ερώτημα. Ποια είναι η νομική βάση σας για να δράσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ψάξαμε, ψάξαμε και μιλήσαμε με ένα σωρό νομικούς παγκοσμίω. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο νόμος που έδωσε το δικαίωμα στα GCHQ και στον νόμο Βασίλειο και την κυβέρνησή του να κάνουν όσα κάνανε. Βρήκαμε μια υπόθεση, αλλά χρειάστηκε να περάσουμε από ειδικό δικαστήριο για έρευνες, ένα δικαστήριο ε, ιδιαίτερο και μυστικό το οποίο ε, ουσιαστικά ε, το έργο τη κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν θέλω να τον να κάνω ενεργητικού υπενιχμού για τη λειτουργία του δικαστηρίου, αλλά την, το έχει καταρτήσει η ίδια η GCHQ. <laughs> το δεύτερο είδο δράση ε, είναι αυτό που μόλι την περασμένη εβδομάδα έγινε, ω προ το τέμπορα πάλι, αλλά έχει να κάνει με τη σχέση με τι εταιρείε. Επικεντρωθήκαμε εδώ παρανόμω, με τις, ε, μάλλον ε, επικεντρωθήκαμε κακώς στις εταιρείες που, ασχολ, που ενεπλέξαν στο πρίσμ. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι έγινε και με τις εταιρείε που πήραν μέρος στην παρακολούθηση των υποθαλάσσιων καλωδίων. Αποστήλαμε επιστολές στον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, διότι όσα εργάζεται επί της, ε, του σεβασμού των εταιριών ως προς τις απαιτήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, εδώ εμπλέκονται η BT, η Verizon UK, η Vodafone Cable, η Level 3, η Viatel. Όλοι αυτοί είχαν δώσει πρόσβαση στα καλώδια τους. Εδώ ε, απλώς ρωτήσαμε τις εταιρείες αυτές. Πότε σας ζητήθηκε από την GCHQ να δώσετε πρόσβαση στα υποθαλάσσια καλώδια σας. Τι κάνατε όταν σας το ζητήσαν αυτό. Σας ζητήσατε την νομική βάση, αντισταθήκατε, Αναζητήσατε άλλε νομικέ εναλλακτικέ, νόμιμε, μάλλον εναλλακτικέ. Και ποιε είναι οι πολιτικέ σα αντιδράσει όταν δέχεστε μια κυβέρνηση από οπουδήποτε μέρο του κόσμου για να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σα, των οποίων όμω δεν είστε κάτοχοι εσεί, απλώ τα διαθέτετε για ένα χρονομενό διάστημα. Όπω η Level 3 Google, οι οποίοι μπορούν να δώσουν ε, κατάλογο για τους ε, παροχέ τη Google ανά τον κόσμο κατάλογο των καλωδίων της Google. Ε, ας επανέλθουμε όμως στο θέμα του απορρίτου και της εποπτείας. Αυτό που θέλουμε να συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες χώρες είναι ότι ακόμη και για το απλό θέμα της εποπτείας, εποπτείας από κοινοβουλευτικές επιτροπές, ε, τι μπορεί να γνωρίζει μια κυβέρνηση το πραγματικό ερώτημα. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν ε, μονοπόλιο για τη γνώση του τι ακριβώς πράττουν. Όπως είπε και ένας ε, γερουσιαστής στις Ηνωμένες στην επιτροπή ε, που ήταν υπεύθυνη για τα θέματα εποπτείας. Μιλάμε για το παιχνίδι με τις 20 ερωτήσεις. Δεν ξέρει κανείς ποιες ερωτήσεις να θέσει. Ποιος θα σκεφτόταν να ρωτήσει «Έχετε παραβεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας» Κανείς δεν θα σκεφτόταν να θέσει ένα τέτοιο ερώτημα στο διευθυντή ενό φορέα, οργανισμού μάλλον, μια μυστική υπηρεσία. Η νομοθεσία είναι έτσι διατυπωμένη, ώστε το κοινοβούλιο δεν έχει στην ουσία καμία εποπτεία καμία δυνατότητα ελέγχου. Ακόμα λιγότερο κοινοβουλευτική επιτροπή. Για παράδειγμα, ο νόμος του 1984 για τις τηλεπικοινωνίες δίνει δικαίωμα στον ε, Υπουργό να ε, διατάξει εταιρεία τηλεπικοινωνίας να συμμορφωθεί με κάποια εντολή. Η εντολή αυτή μπορεί να είναι οποιοδήποτε περιεχομένο. Οι εντολές όμως αυτές, οι αποφάσεις αυτές μπορεί να μην ε, παρουσιαστούν στο κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο μπορεί να τις αγνοεί. Υπήρξε έφεση το 2000 με ε, τον κανονισμό για τις ερευνητικές αρμοδιότητες. Και πρόσφατα μιλήσαμε για τον νόμο που προτάθηκε το 2012 για τα δεδομένα των επικοινωνιών. Η ιδέα που υποκρύπτει το νομοσχέδιο αυτό είναι ότι οποιοδήποτε παροχέας στο Ηνωμένο Βασίλειο παράσχει ε, τηλεπικοινωνίες δεν μπορεί να με τα δεδομένα, οποιοδήποτε χρήστη ε, πολίτη που βρίσκεται εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου χωρί να το γνωρίζει το Κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα νομοθετήματα έχουν να κάνουν με λευκέ νομοθετικέ επιταγέ που ουσιαστικά ε, αποδίδονται ε, στι μυστικέ υπηρεσίε. υπηρεσίες. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν ό,τι έρευνα θέλουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να γνωρίζει το κοινοβούλιο τίποτα για το τι δράση αναλαμβάνεται. Ούτε καν αν αυτό επιτρέπεται ή είναι εφικτό. Οπότε ξαναρωτώ, οποιοδήποτε κοινοβούλιο να ε, αναμένεται να γνωρίζει τι ερωτήματα πρέπει ποιο είναι το εύρο των μυστικών προγραμμάτων, τι ερωτήσει πρέπει να θέσει. Μάλλον δεν εκπλήσει κανέναν που ιδιαίτερα στι ΗΠΑ και το ΗΠΑ οι ε, ε, επιτροπέ εποπτεία των ε, μυστικών υπηρεσιών στο μεγαλύτερο μέρο είναι σαν μαζορέτε. Μαζορέτε που επιθυμούν υπέρ των μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή ξέρουν πολύ λιγότερα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους από τις ίδιες οι μυστικές υπηρεσίες. Αυτό αποδεικνύεται από την περασμένη εβδομάδα ανακαλύψαμε ότι στη Βουλή των Ορδών έγινε συζήτηση για τα προγράμματα αυτά. Και υπήρξε διαρροή όταν ένα μέλο τη ε, Επιτροπή Αποκτίας των Μυστικών Υπηρεσιών και πριν από τι αποκαλύψει Νόντεν είπε ότι πριν από τι αποκαλύψει μάλλον αυτέ η Επιτροπή ουδέποτε είχε συζητήσει το πρόγραμμα PRISM. Μόνον μετά τι αποκαλύψει του Σνόντεν. Δεν το γνώριζαν δεν ήξεραν τι μπορούν να ρωτήσουν εάν η κυβέρνηση μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Google, εάν η κυβέρνηση μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τη Microsoft. Δεν ήξεραν τι ερωτήσει να ρωτήσουν. Όταν έσκασε η βόμβα του Snowden, τότε καταλάβαν ότι κάποια σχέση έχει με όλα αυτά τη GCHQ. Πρόσφατα ένα πρώην μέλο τη κυβέρνηση και πρώην μέλο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλεία έγραψε στην Guardian, ανέφερε στην Guardian, ότι σε μία διετία κανένα από τα μέλη της Επιτροπής δεν ήξερε για το πρόγραμμα Τεμπόρα, ούτε καν είχε συζητηθεί. Είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα. Εάν σκεφτείτε τι γίνεται με την εκτελεστική λοιπόν εξουσία, δεν μπορούσε να συζητήσουν το πρόγραμμα Τεμπόρα, δεν το γνώριζαν. Δεν μιλάμε για τους απλούς πολίτες όμως. Εάν σκεφτείτε λοιπόν τον νόμο για τις επικοινωνίες που συζητήθηκε προηγουμένως, και δείτε τι γίνεται. Αυτά είναι παραδείγματα του πώς, πώς ήταν καθοριστικής σημασίας, πώς μάλλον η όλη προσπάθεια εποπτείας έχει παρακαμφθεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ζήτησε το 2008 από την GCHQ να συγκεντρώνει δεδομένο οποιοδήποτε χρήστη του διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Αυτό θεωρήθηκε παράδειγμα, Οπότε εγκαταλείφθηκε αυτή η πολιτική. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Τα δεδομένα επικοινωνία ε, πάλι εισήχθησαν το 2012, όχι όμω σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Και το Κοινοβούλιο έκανε μια συζήτηση για το κατά πόσον επιτρέπεται αυτό για τα μεταδεδομένα. Αλλά επί τη ουσία τα βασικά στοιχεία, τα μεταδεδομένα υπήρχαν και η GCHQ τα ε, συγκέντρωνε. Ακόμη και το 2012 όταν είχε απορριφθεί από το Κοινοβούλιο σχετική πρόταση. Να ολοκληρώσω λέγοντα και προβλέποντα ποια είναι η μελλοντική μα πορεία. Όπω είπε ο κ. Μπίκφορντ, θα πρέπει να προβλέψουμε και άλλε εγγύησει για τι διαδικασίε, όπω ε, ε, διαδικασίε ε, έγκριση με την επιβολή του κράτου δικαίου. Αυτέ οι υπηρεσίε, οι μυστικέ υπηρεσίε λειτουργούν εδώ και χρόνια χωρί επαρκή ελέγχου και τώρα είδαμε τι γίνεται όταν υπάρχουν έλεγχοι. Χρειάζεται λοιπόν να ολοκληρωθεί η εποπτεία γιατί βλέπουμε ότι το μέχρι τώρα μοντέλο μας έχει ε, αποτύχει και χρειάζεται ε, αναθεώρηση. Πρέπει να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση. Ποιε είναι οι αρχέ που ε, διέπουν την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μοντέλα εποπτείας. Οι οργανώσει πολιτών ανά τον κόσμο και πολλοί ειδικοί ανά τον κόσμο συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν τα τελευταία χρόνια αρκετέ φορέ προκειμένου να εκπονήσουν κάποιε συγκεκριμένε αρχέ για το πώ πρέπει να γίνεται η εποπτεία των προσωπικών δεδομένων και σε συμφωνία με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι 13 από τι αρχέ απεστάλησαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Σουηδία τον περασμένο μόλι μήνα μίλησε για την ανάγκη να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση για τα θέματα αυτά. Η πρότασή μα είναι αρκετά μετριοπαθή και ταπεινή. Δηλαδή, χρειάζεται ισχυρότερο ε, νομοθετικό πλαίσιο για την δημοκρατική εποπτεία. Θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικοί νόμοι που να επιτρέπουν την εποπτεία από την κυβέρνηση και να την διέπουν. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις, να υπάρχουν συγκεκριμένοι νομικοί στόχοι για την εποπτεία με συγκεκριμένους ορισμούς όρων όπως η εθνική ασφάλεια ε, και η οικονομική ευημερία, ειδικά για το Βασίλειο. Η εποπτεία πρέπει να είναι δεσμευτική και αναγκαία και οι παρεμβάσει πρέπει να, είναι, ε, να βασίζονται στην αρχή τη αναλογικότητα. Πρέπει να χρειάζεται δικαστική έγκριση και απόφαση και η δίκαιη διεξαγωγή των διαδικασιών θα πρέπει να βασίζεται στην μη απόρριτη ε, ανταλλαγή πληροφοριών και τι σχετικέ συμφωνίε. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση των ατόμων που ε, παρακολουθούνται και Επίση, να μην ε, ξεπούνται όλα τα παραθυράκια που μπορεί να επιτρέπει το κράτο δικαίου. Αυτέ δεν είναι τυχαίες ιδέες, είναι στοιχεία που έχουν συζητηθεί ανά την ε, Ευρώπη, επίσης στη διεθνό, στο διεθνές δίκαιο, σε περιπτώσεις παρακολούθησης, εποπτείας και <clears throat> τήρησης των δικαιωμάτων. Έτσι θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε την πορεία μας προς μια κοινωνία σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιοσύνης. Μόνο εφόσον αυτοί οι κανόνες τηρηθούν θα μπορούμε να ξανασυζητήσουμε για το θέμα της εποπτείας. Την εποπτεία μπορούμε να την προβλέψουμε όταν αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου. Η εποπτεία θα πρέπει να διατηρεί και να προστατεύει το κράτος δικαίου, όχι αυτό που κάνει τώρα, να παίζει το ρόλο μιας εθνικής ε, μαζορέτας που επικροτεί την εποπτεία. Ευχαριστούμε. Τώρα οι ερωταπαντήσει. Καταρχήν η Σκιώδη, ο κύριο Κοέλιο θέλει να θέσει ερώτημα, εξ του Άξελ από το ΕΛΚ που δεν μπορεί να προσέλθει. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ Κλάβιε. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του κύριου Μπίκφορντ που τόνισε την ανάγκη δικαστικής εποπτείας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της χώρας μου όπου κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να επιτρέψει την υποκλοπή επικοινωνιών. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλοί υπουργοί έχουν τη δικαιοδοσία να το πράξουν και συμφωνώ ότι δεν αρκεί η δικαστική εποπτεία ex post factum, facto. Και αυτό όχι μόνο γιατί γίνεται μετά κατόπιν εορτής, αλλά και γιατί, από ό,τι ξέρω, μόνο ένα μικρό μέρος των επιτηρήσεων γίνονται γνωστές. Οι περισσότερες αγνοούνται. Δεν συμφωνώ λοιπόν, ε, συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας. Και συμφωνώ και με τον κύριο Έλσεν που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η εποπτεία αλλά η τήρηση του νόμου. Αλλά μια καλή εποπτεία είναι ουσιώδης για να σε γίνει σεβαστός ο νόμος και θα ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο, να σας ζητήσω να μου εξηγήσετε πρώτον για την κοινοβουλευτική εποπτεία. Πώς μπορεί να υπάρξει μια σωστή τι αυτή αν τα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν οριστεί από τον Πρωθυπουργό και δεν έχουν εκλεγεί από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει στον Ηνωμένο Κοινοβούλιο μία επιτροπή τέτοια που όρισε ως πρόεδρο έναν από το κόμμα της αντιπολίτευσης αλλά μπορεί να υπάρξει πραγματική κοινοβουλευτική εποπτεία με τέτοιες παρεμβάσεις επίσης για τη δικαστική εποπτεία μου έχουν πει ότι στο ΙΤΑΒ οι δικαστές έχουν το δικαίωμα να κρίνουν ex post facto πράξεις. Υπάρχει εδώ σωστή εποπτεία. Ευχαριστώ πολύ. Uh, but um, it's just a British conversation here. Um, just um, colleagues, there will καμιά σύντομη απαντησούλα στον κύριο Κοέλιο. Πρώτα ο Δαβίδ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλές ερωτήσεις, ιδιαίτερα από τον Γάλλο βουλευτή. Το σύστημα δικαστικής εποπτείας με επικεφαλή στον αρμόδιο δικαστή λειτουργεί πολύ καλά, αλλά η ex post facto ίσως δεν λειτουργεί τόσο καλά. Πρέπει να αρχίσουμε όμως από το εξή. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, μάλλον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια ότι η συλλογή πληροφοριών είναι κάτι πολύ δύσκολο και δύσκολο επίσης είναι να το χειριστούμε σωστά, να το ρυθμίσουμε σωστά γιατί μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι εάν υπάρχουν οι νόμοι και όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται ως προς την αναγκαιότητα της δράσης και την αναλογικότητά τους γίνεται με επαρκή εποπτεία, τότε μπορούν οι μυστικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν όσο ελεύθερα πρέπει να λειτουργήσουν για να προστατέψουν το κοινό. Αλλά με επαρκή εποπτεία και άρα να μην γίνεται κατάχρηση. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα. Η κοινοβουλευτική επαπτεία δεν λειτουργεί ούτε και ούτε και οι δικαστικές έρευνες που γίνονται κατόπιν εορτής πολλές φορές πολύ αργότερα και μόνο επιλεκτική μπορεί να είναι αν θέλουμε σωστή εποπτεία τότε πρέπει να έχουμε δικαστή για να εξισορροπήσει να κρίνει την ομιμότητα των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Εκείνος είναι ο εξισορροπητής ή εκείνη και είναι πολύ σημαντικό αυτό διότι αν υπάρχει τέτοια εξισορρόπηση τότε μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος καταχρήσεων και επομένως από εκεί και πέρα ό,τι εποπτεία θέλετε από κοινοβουλευτικούς που να τους έχουν ορίσει άλλοι κοινοβουλευτικοί, μέλη δικαστηρίων που επίσης να τους έχουν ορίσει κοινοβουλευτικοί και όχι ο Πρωθυπουργό. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μειώνουμε τον κίνδυνο γιατί ποτέ δεν θα είναι τέλεια τα πράγματα αλλά αυτό που θέλουμε είναι να μειώσουμε τον κίνδυνο καταχρήσεων στο ελάχιστο δυνατόν. Και νομίζω ότι το γαλλικό σύστημα με με ένα δεύτερο βοηθητικό ανεξάρτητο σύστημα θα επέτρεπε στις μυστικές υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους και να μας προστατεύουν αλλά επίσης να μειώνεται το περιθώριο καταχρήσεων. Στο ΙΤΑΒ τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι είπατε. Τώρα προεδρεύει της Ερευνητικής Επιτροπής ένας πρώην Πρωθυπουργός που είχε λάβει μέρος σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αλλά τις έχουν δοθεί και πρόσθετες δικαιοδοσίες που μπορεί να είναι ανεπαρκείς αλλά είναι πολύ περήφανοι για αυτές. Και ο νόμος επιτρέπει στο εκτελεστικό να κατακρατά πληροφορίες και από τέτοιε επιτροπές. Πώς μπορεί να υπάρχει λοιπόν εποπτεία άμα δεν δίνεται πρόσβαση στην πληροφόρηση. Το άλλο για την Κομισιόν όχι για την Επιτροπή Δικαστών. Ο αρμόδιος δικαστής δεν είναι ανάγκη να είναι τρέχον δικαστής, μπορεί να είναι πρώην δικαστής. Υπάρχει ένα γραφιάκι που διεκπεραιώνει όλες τις ε, τεχνικές αιτήσει για έρευνες. Ε, δεν προλαβαίνει λοιπόν. Η κοινοβουλευτική εποπτεία γενικότερα και το, αυτό που εξηγεί γιατί η κατάσταση είναι τόσο άσκημη στο ΙΤΑΒ είναι ότι μπορεί να μην γνώριζαν για τα προγράμματα μυστικής παρακολούθησης αλλά και να τα γνώριζαν ε, είτε τα γνώριζαν είτε δεν τα γνώριζαν παρόλα αυτά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Επάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Κοέλιο να συνεχίσω. Σε σένα Δαβίδ. Για αυτό το θέμα των εντολών των πολιτικών κάποιος το MI5 ή το MI6 που μπορεί να είχε λειτουργήσει σε διευθυντική θέση θεωρούν τα κόμματα ότι δεν θα ήταν σωστό να προεδρεύει σε τέτοιου είδους έρευνες όπως έχει γίνει και με υπουργού εσωτερικών. Και αυτά δεν έχουν αλλάξει. Η κατάσταση λοιπόν δεν έχει καθόλου εξυγχρονιστεί. Λες τώρα για το γαλλικό σύστημα με επικεφαλής δικαστάς. Ερωτώ λοιπόν, γιατί σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε και μερικές συστάσεις και να δούμε σε τι νομικό πλαίσιο θα, γίνεται, θα γινόταν καλύτερα η υποπτία. Ερωτώ λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ότι δεν έχουμε αλλάξει τα πράγματα, δεν έχουμε βάλει επικεφαλής δικαστάς και τα αφήσαμε όλα όπως ήταν. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένο. Ο καθηγητής Κάμερον μας είπε ότι το γερμανικό και σουηδικό σύστημα είναι πιο εύκαμπτο, είναι πιο μικρέων διαστάσεων η υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών. Ίσως και αυτό είναι λάθος στο έγγραφό μας. Το δικό μας σύστημα συγκριτικά δεν είναι τόσο ευέλικτο. Μήπως υπάρχει ένα διαρθρωτικό λοιπόν πρόβλημα και όχι μόνο πολιτικό. Εσύ είχες υπάρξει νομικός σύμβουλος ή διευθυντής μάλλον στο MI5. Η πολιτική δεν πρόκειται να δεχτούν να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους. Μήπως γι' αυτό δεν αναμορφώθηκε το σύστημα. Τι φρονείς. Μία από τις μυστικές υπηρεσίες μας ε, έχει κατηγορηθεί για τέτοιου είδους καταχρήσεις. Πολύ καλό ερώτημα, σας κατευχαριστώ. Καταρχάς, η ακαιρεότητα των υπηρεσιών και των υπουργών δεν τίθεται σε αμφιβολία. Έχω συνεργαστεί μαζί τους σε πολλά, πολλά χρόνια και η ανομαλία που υπάρχει είναι ότι υποφέρουν οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών γιατί είναι αναγκασμένοι να ψεύδονται προς το κοινό αλλά αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλειά του. Έχουν λοιπόν μεγάλη ακαιρεότητα και αυτό είναι και το κυριότερο κριτήριο όταν προσλαμβάνονται. Τώρα για τους υπουργούς σε σύγκριση με τους δικαστάς. Από ό,τι ξέρω εγώ, λόγω της υπόθεσης Λεάνδρου, δεν μπορούμε να πούμε, να καταλάβουμε τα πράγματα, εκτός αν επανέλθουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάσουμε τη σύμβαση και δούμε τι εξισορροπήσεις προβλέπονται εκεί. Η υπόθεση Λεάνδρου ήταν προφανής, διότι φάνηκε από εκεί ότι η αναγκαιότητα μιας παρέμβασης και η αναλογικότητα είχαν γίνει σεβαστές με την ηλεκτρονική παρακολούθηση τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η τεράστια αυτή δραστηριότητα ε, δεν παρακολουθήθηκε όπως έπρεπε από τους κοινοβουλευτικούς γιατί δεν προλάβαιναν να την παρακολουθήσουν. Το θέμα είναι να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Αλλά τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο καταλάβαμε ξαφνικά ότι αν έχουμε 13 βασικές αρχές και αυτά που μας είπε ο καθηγητής Κάμερον θα πνίξουμε την λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας προστατεύουν πια τόσο αποτελεσματικά. Άρα χρειάζεται μια πιο συμπυκνωμένη, πιο ευέλικτη παρακολούθηση, η εποπτεία. Και εδώ γι' αυτό επανέρχομαι στο γαλλικό πρότυπο. Αν υπάρχει ο δικαστής που συνεργάζεται με τις μυστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της διενέργειας μιας έρευνας, τότε παίζει ένα ρόλο ανεξάρτητο και όχι πολιτικό. Και έτσι είναι, αυτή είναι η καλύτερη δυνατότητα που έχουμε για να εξισορροπήσουμε αναλογικότητα και ανάγκη για να μην υπάρξει κατάχρηση και επίθεση στην ε, ιδιωτική ζωή των πολιτών. Πολύ σωστά νομίζω ο καθηγητής εδώ κατέκρινε το, το Βρετανικό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τέτοιες έρευνες δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση κλάς και θα πει δεν μπορούμε πια να δεχθόμαστε εποπτεία από βουλευτάς. Χρειάζεται δικαστική. Και υποψιάζομαι ότι και εκείνοι θα επιλέξουν το γαλλικό σύστημα. Ωραία. Επόμενη ερώτηση από τον Γιάνν Αλμπραχτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που ήρθατε ε, και είστε ενώπιον μας. Χρειαζόμαστε την εμπειρία σας και την πραγματογνωμοσύνη σας και εμείς Επιτρέψτε μου να πω ευθύ εξ αρχή. ότι χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή ακριβώς τη μέρα γίνεται έλεγχο και στη Βουλή των Κοινοτήτων, στο Ηνωμένο ναι. Βασίλειο. Ας ελπίσουμε να κινηθούν και τα εθνικά κοινοβούλια και του Ηνωμένου Βασιλείου εμπροκειμένου. Πρέπει όμως να σας πω ειλικρινά ότι κατά την άποψή μου υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έργο που καλούμεθα εμείς να φέρουμε σε πέρας. Και είναι το εξής. Όλα αυτά που γίνονται στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες συνάδουν με τις αρχές τις οποίες συμφωνήσαμε. Και βλέπω αυτό που είπατε για το CCHR, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά Υπάρχει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι δεσμευτικός και για το Ηνωμένο Βασίλειο στη συνθήκη της Λισαβόνα. Θα πρέπει να εργαστούμε λοιπόν ε, προς την κατεύθυνση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που ήρθατε να τα συζητήσετε μαζί μας. Έχω μια ερώτηση πρώτα για την, ε, το νόμο ΡΥΠΑ. Δηλαδή ποια είναι η νομική βάση στο α4 για το πρόγραμμα Τέμπορα. Θα μπορούσατε λίγο να επεκταθείτε σε αυτό. Τι γίνεται όταν υπάρχει ένα ένταλμα για το 8-4 γιατί στο ιστορικό του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ορίζεται ρητά το πεδίο εφαρμογής ή το πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται αυτή η παρακολούθηση. Δεν μπορεί να αφορά ένα ε, καλώδιο οπτικών ινών υποβρύχιο κιόλα. Πρόκειται για συγκεκριμένο πεδίο ή συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν σου λέει το έντολμα να πας να παρακολουθήσεις τα καλώδια. Και αυτή η εντολή υπουργική συνοδεύεται από κάποιο πιστοποιητικό του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών ή ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία συστημάτων και προγραμμάτων τύπου τεμπόρα. Γιατί τελικά αυτό έχει να κάνει και με την κατασκοπία ή την ανάλυση ε, δεδομένων εκτός της επικράτειας ή που προέρχονται από ε, την αλλοδαπή. Και πού μπαίνει η εθνική ασφάλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν πρόκειται για την κοινή μας ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρώτο ο Ντέιβιτ και μετά ο Γκάς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία για το τέμπορα και το ρήπα. Η απάντηση είναι η εξή. Το δικαστήριο το αρμόδιο για τις ερευνητικές εξουσίες θα αποφανθεί μετά την καταγγελία σε πρώτο λόγο και σε δεύτερο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Mm. Μέχρι εκεί μπορώ να σας απαντήσω για αυτό το θέμα. Για το Υπουργείο Εξωτερικών ή μάλλον ε, υφυπουργοί ε, και μυστικές υπηρεσίες αλλά και αστυνομία και ιδιοκτικές αρχές σε υψηλό επίπεδο μπορούν να αποφασίσουν για το αν θα υπάρξει μυστική παρακολούθηση ή όχι. Ο Γκάς, Περιγράψατε ακριβώς την περίπτωση που μας αφορά. Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται και ακριβώς αυτές τις ερωτήσεις κάνουμε και εμείς ε, για τα πιστοποιητικά και τα εντάλματα. Κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ε, η κοινότητα αυτή των υπηρεσιών πληροφοριών απαντώντας τις αποκαλύψεις για το πρίσμα και το τέμπορα τι έκαναν. Αμφισβήτησαν το νομικό πλαίσιο για το κατά πόσο τα δάλματα ρήπα και ο νόμος για τις μυστικές υπηρεσίες του 1994 ε, μπορεί να καταργηθεί από το νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εμείς έχουμε απευθυνθεί προδικαστικά στο αρμόδιο δικαστήριο για το ερώτημα. Όλα αυτά όμως που καταλήγουν. Ε, στη υπόθεση αυτή αρχής είναι σωστό μια κυβέρνηση να κάνει διάκριση μεταξύ των εγχωρίων επικοινωνιών και των λοδαπών. δηλαδή μεταξύ Αμερικανών και μη Αμερικανών, μεταξύ αλλοδαπών και πολιτών της χώρας. Είναι παγκόσμια επικοινωνία σήμερα και η οικονομία και δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τέτοια διάκριση. Και όλη η ιστορία του ε, ρέπα αυτού ε, του θέματος με τα εντάλματα είναι να διατηρηθεί η ε, διάκριση μεταξύ του εμείς και του εσείς. Η Κορνέλια, ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη διάκριση Αμερικανών και μη ε, το έχουμε ξαναζήσει και το είδαμε και στο ταξίδι μας στην Ουάσιγκτον. Σας ευχαριστώ πολύ αυτά που μας είπατε. η κατάσταση είναι αυτή που είναι και η μέρα γκρίζα και η ζωφερή σήμερα δεν μας γεμίζει αισιοδοξία. Αλλά τι να κάνουμε. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Ρωτήσατε για τη νομική βάση. Για όλα αυτά την ψάξατε και δεν βρήκατε νομική βάση. Και αν υπάρχει κάποια για ε, αυτή τη μαζική παρακολούθηση, είπατε ότι είναι κάποιοι χαλαροί νόμοι και ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει πραγματική εποπτεία, σου λένε ότι είναι απόρριτα αυτά, μας εξαπατούν κιόλα. γιατί να μην το πούμε ξεκάθαρα, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και είπατε ότι πρέπει να ενισχυθεί η νομική βάση και να επανέλθει το κράτο δικαίου. Και ρωτώ, πού θα πρέπει να γίνει η αρχή εκεί πέρα. Και τι συστάσεις θα κάνετε και προς ποιους. Για να επανακατασταθεί, να αποκατασταθεί μάλλον η ε, ισχύ του κράτους δικαίου, όπως το είπατε. Και κάποια στιγμή καταλήγουμε στον πολίτη, ε, άντρα ή γυναίκα, που είναι εκτεθειμένη και έρμεο απέναντι στην κατάσταση αυτή. Αυτούς πώς θα τους ε, αντιμετωπίσουμε και τι μας συστήνεται για να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη προστασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει, ο προστάτευτος πολίτης. Και όλα αυτά που ακούμε δεν είναι πολύ αισιόδοξα και λογικό και επόμενο είναι. Τι μας συνιστάτε. Και ένα τρίτο, όπως γνωρίζετε, στη Γερμανία έχουμε την Εξεταστική Επιτροπή για το, την υπόθεση NSU και έχουμε περισσότερα προβλήματα με τις μυστικές υπηρεσίες, την υπηρεσία προστασίας του συντάγματος. Όχι ότι παρακολουθεί, αλλά τι παρακολουθεί. Γιατί εκτίμησε πάρα πολύ λάθος πράγματα ε, ως απειλή, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν απειλή. Και αυτά που ήταν απειλή και έπρεπε να τα παρακολουθούσαν, τους ξέφυγαν. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι μόνο η αναλογικότητα και ε, η ισορροπία, αλλά το τι συνιστά απειλή και πώς αξιολογείται κάτι ως απειλή για να το αντιμετωπίσεις και να συλλέγεις στοιχεία. Όχι μόνο ότι παρακολουθείς και ποιον παρακολουθείς, αλλά για ποιο λόγο τον παρακολουθείς και τι δεν ε, καταγράφεις. Όλα αυτά είναι προβλήματα. και ε, Θα ήθελα να ακολουθήσω την, να ακούσω συγγνώμη, την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κορνίλια. Ο Ντέιβιτ και μετά ο Γκάς. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω πολύ περισσότερο προς τις συστάσεις και το πώς βλέπω το μέλλον σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, βεβαίως, αυτά θα πρέπει να τα ορίσουν οι αναλύσεις των μυστικών πληροφοριών από τις ίδιες τις μυστικές υπηρεσίες. Το τι θα γίνει έπειτα για τον κίνδυνο είναι κάτι που εκείνοι πρέπει να το ζητήσουν, βάσει της προτασής μου, από τον ε, ανακριτή επιτόπου για το τι πληροφορίες πρέπει να αποκαλύψουν τι πληροφοριότητε πρέπει να χρησιμοποιούν και μετά ο δικαστή θα αποτιμήσει τα δικαιώματα του ενόμου ε, προσώπου και τις δράσεις της υπηρεσίας. Μετά θα λυθεί η απόφαση, κατόπιν της εξέτασης αυτών των δύο σκελών. Χρειάζεται ένας νόμος συνολικά για την εποπτεία. Ως τώρα, σε πολλές χώρες υπάρχει ένα συνοφίλευμα αρμοδιοτήτων κυβερνητικών και Υπάρχει νόμος για τις μυστικές υπηρεσίες, για τις επικοινωνίες, ε, την πρόσβαση στις πληροφορίες διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την κράτηση των δεδομένων, διότι η κυβέρνηση το ήθελε αυτό επίσης. Πρέπει να σταματήσουμε να νομοθετούμε αναλόγω με το τι θέλουν οι μεστικέ υπηρεσίε και να ζητήσουμε ένα συνολικό νομικό πλαίσιο. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη μαζική παρακολούθηση ταυτόχρονα όμω. Δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει κανείς να ερευνήσει το κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιούνται και να πραδιάζονται οι τεχνολογικέ ε, δυνατότητε, Τα πρωτόκολλα ασφαλεία, τα διάφορα πρότυπα. Είναι απίστευτη η δράση των μυστικών υπηρεσιών που ε, χειρίζονται όπω θέλουν τα πρωτόκολλα τα οποία όλοι απαιτούμε προκειμένου να υπάρξουν εμπορικέ συναλλαγές τα οποία χρειάζονται για τι καθημερινές μα υποθέσει. Και επίσης ε, είμαι αισιόδοξο για να πω την αλήθεια. Πραγματικά είμαι αισιόδοξο. Τα πράγματα θα βελτιωθούν. Διότι ενώ η GCHQ έκανε ό,τι ήθελε παλιότερα τότε που το έλεγε και Telegraph, ε, ότι οι κυβερνήσεις ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν τον τηλέγραφο κάποτε. Οι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο οι ίδιοι, επικοινωνούν οι ίδιοι διακρατικώς. Οι εταιρείε φροντίζουν να υπάρχει εμπιστοσύνη από την πλευρά των πελατών, των καταναλωτών, ότι μπορούν να επικοινωνούν και να γράφουν ένα στον άλλο σε συνθήκες ασφάλειας. Γι' αυτό το τέμπερο είναι σημαντικό. Γι' αυτό μια σχετική δύναμη κρούσης είναι σημαντική. Γι' αυτό είναι σημαντική η μηχανική. Οι εταιρείε είναι σημαντικέ. Θα θυμώσουν πάρα πολύ όταν καταλάβουν τι είδου παραβιάσει μπορούν να υπάρχουν στα συστήματα για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι. Πρέπει να μπορούν να μα έχουν εμπιστοσύνη. Πολύ σύντομη παρατήρηση. Μην ξεχνάμε ότι οι τρομοκράτες οι ομάδε οργανωμένου εγκλήματο έχουν πρόσβαση σε προηγμένα μέσα και εκείνοι, προηγμένα μέσα επικοινωνίας, το σκοτεινό δίκτυο, όπως λέγεται, dark web και ούτω καθεξής, άλλες προηγμένες μεθόδους. Επίσης, πολλοί προηγμένες μεθόδους ε, hacking, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα απόρριτα και των κυβερνήσεων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και να καταλάβουμε ότι κάποιε φορέ όντω πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο τη εποπτεία, αλλά να αντιμετωπίζονται και αυτέ οι απειλέ. Ιδάλλως μπορεί να διατρέχουμε και κίνδυνο. Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση. Η κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ. Είπατε ότι εδώ πρέπει να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου, κύριε Χώσεκ πριν η εποπτεία αποκατασταθεί με τη σειρά της. Νομίζω ότι δεν είναι απλώς το κράτος δικαίου, αλλά η ίδια η δημοκρατία. Για τη δημοκρατία μιλάμε. Διότι αυτό που αισθάνομαι είναι ότι μπορεί να υπάρχουν διαστροφές της δημοκρατίας, πραξικόπημα που εν εάν δεν βεβαιωθούμε ότι θα επιστρέψουμε στο κρατό δικαίου και ότι όντω θα λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα και η δημοκρατική εποπτεία. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Ξεκινώντα από τι ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, όταν επισκεφτήκαμε τι ΗΠΑ, ρώτησα τον Μάικ Ρότζερ, ένα γερουσιαστή που είναι και πρόεδρο τη ε, Επιτροπή τη Γερουσία για την εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών, ρώτησα αν δεν το ξέρε ο πρόεδρο, ποιο το ξέρε. Το ξέρει η Επιτροπή. Δεν απήντησε. Δεν ξέρω λοιπόν αν είχε γνώση, αν δεν ήθελε να το πει ή αν δεν γνώριζε. Και ούτε αυτό ήθελε να το πει. Τι σημαίνει αυτό. ο Big Brother έχει ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Από κάθε έλεγχο. Γι' αυτό ρώτησα πολλού από τους παρε, Τι θα γίνει μετά. Κατασκοπία κατά του Πρόεδρου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και ποιο είναι το ερώτημά σας, Άννα. Έρχεται. Ναι, στην περίπτωση της Βρετανίας. Ας το συσχετίσουμε με αυτό. Κύριε Μπίγκφορντ, είπατε ότι ο πρόεδρος Μπούς ε, παρέκαμψε την αποψηφίζα. Οι οποίοι αποδυναμώθηκαν έτσι περαιτέρω. Μπορείτε να μας πείτε, αν υπάρχει κανείς, κάποιος που να γνωρίζετε, που να συνελήφθη, λόγω ακριβώς αυτής της παράκαμψης. Κάποιος που να έπαθε κάτι. Αυτός, αυτή η χειραγώγηση των υπαρχόντων μηχανισμών προκάλεσε κάποιο θύμα. Και σκεφτείτε λίγο τη συνεργασία που υπάρχει με την Βρετανία. Εφόσον υπήρξε συνεργασία με τη Βρετανία. Το ερώτημα μου είναι πώς η Βρετανία με τη σειρά τη στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ πώς συνεργάζεται με ένα σύστημα που είναι ανεξέλεγκτο. Δεν μιλάω για το Βρετανικό, μιλάω για το Αμερικανικό. Και έπειτα, για το Βρετανικό σύστημα. Να υποθέτουμε ότι εάν υπάρξει ανάγκη λόγω χάρη ο Βελγικός Φορέας Τηλεπικοινωνιών. Εάν η Belgacom λοιπόν, η εταιρεία, δεχτεί επίθεση από hacker, από την GCHQ συγκεκριμένα, θα μπορούσε να έχει δώσει την εντολή ένας ε, Βρετανός Υπουργός και αν αποδειχτεί ότι η Βρετανική Πρεσβεία στο Βερολίνο αστεί κατασκοπία από τη στέγη του κτηρίου αυτό μπορεί να γίνεται εν γνώση κάποιου Βρετανού Υπουργού ή με την εντολή του να υποθέσουμε τέτοια σενάρια. Και στη Βρετανία υπάρχει κάποιο όριο που όλα αυτά να σταματούν. Ή είναι όλα ανεξέλεγκτα όπως συμβαίνει προς στιγμή στις ΗΠΑ. Και επίσης να ρωτήσω για τη συνεργασία με άλλες μυστικές υπηρεσίες, με άλλους φορείς μάλλον στην Ευρώπη, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Ο κύριος Κουέλιο το είπε. Μίλησα για τη δική μας τη χώρα. Είδαμε πώς το σύστημα μπορεί να γίνει, να παρακαλθεί και να στρεβλωθεί. Τι εμπειρίες έχετε εσείς. Τι παραδείγματα υπάρχει περίπτωση τέτοιες μορφές διεθνούς συνεργασία, όχι μόνο με τι ΗΠΑ, με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς ή εκτός Ευρώπης τέλος πάντων. Υπάρχει περίπτωση κάποιο σύστημα να διασφαλίζει ότι κάποιοι βασικοί κανόνες του κράτους δικαίου τηρούνται, ότι δεν παραβιάζονται. Λόγω χάρη στην περίπτωση εκείνου του Βραζιλιάνου πολίτη που ήταν σύντροφος κάποιου δημοσιογράφου της Guardian Μπορεί να υπήρχε συνεργασία μεταξύ Βρετανικών και Βραζιλιανικών υπηρεσιών. Το ένταλμα σύλληψης το, ζήτησε ο Υπουργός, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο επικεφαλής μιας μυστικής υπηρεσίας, ένας δικαστής. Ποιος? sure δεν είμαι βέβαιο ότι υπάρχουν αυτέ οι απαντήσει από του ομιλητές μα. αλλά θες να δοκιμάσει. Ήταν εκτεταμένη η ερώτηση, είναι πεντάπτυχη. Και ίσω να ολοκλήρωνε κιόλα με κάποιε καταληκτήριες παρατηρήσει αν θέλει. Και οι δυο σα. Για δοκιμάστε με την ερώτηση αυτή και κάποιε παρατηρήσει για να κλείσουμε. Να ολοκληρωθεί αυτό το πάνελ. David. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Άννα. Δεν μπορώ να απαντήσω καμιά από αυτές τις ερωτήσεις. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα γεγονότα. Σε ό,τι φορά το κατά πόσο παρακάμφθηκε το δικαστήριο Φάιζα. Ήταν ε, ένα προεδρικό διάταγμα αυτό που εκδόθηκε. Και υπήρχε και ένας νόμος από το 2008, οπότε το Κογκρέσο ενέκρινε την παράκαμψη του Φάιζα. Ως προς τα υπόλοιπα, όπως είπα και προηγουμένως. Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Ο βαθμός συγκέντρωσης πληροφοριών αυξήθηκε ε, αναλόγως με την αύξηση της απειλής, δηλαδή με τις επιθέσεις από τα άτομα που ε, οι μυστικές υπηρεσίες και οι διοκτικές αρχές ε, ερευνούν. Τα κοινοβούλια να τον κόσμο, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, έχουν ε, καταλάβει ότι όταν χρειάζεται καλύτερη μορφή ελέγχου για την τεράστια άντληση δεδομένων και την σύνταξη προφίλ, συγκεκριμένων προφίλ, θα πρέπει να κάνουν κάτι σύντομα. Δεν πιστεύω ότι η εποπτεία αυτή καθεαυτή πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα παράγοντα που έρχεται να λειτουργήσει εκ των υστέρων. Είναι πολύ αργά όμω τότε. Επίση δεν θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι κανονισμοί ε, θα λύσουν το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα. Ε, υπερβολική ρύθμιση που δεσμεύουν τα εργοτα μυστικών υπηρεσιών και αυτό μας βάζει σε κίνδυνο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να πάμε λίγο πίσω και να δούμε τις βασικές αρχές που διέπουν όλη αυτή τη λειτουργία. Την αναλογικότητα, την αναγκαιότητα και κάποια σχετική σαφήνεια στην νομοθεσία. Αυτά είναι του σημασία. Έπειτα, δικαστική εποπτεία με την συγκεκριμένη γνώση της λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών και υποστηρικτική και εποπτεία από ειδικούς από με υποστηρικτική εποπτεία από τους βουλευτές σε δεύτερη. Δηλαδή να λειτουργούν για την προστασία μας οι μυστικές υπηρεσίες αλλά να υπάρχει και ελάχιστη δυνατότητα καταχρήσεων. Ε, εξαιρετικές ερωτήσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω για την Κομ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λογοδοτήσει μια κυβέρνηση ε, που έκανε επίθεση σε υποδομές άλλης χώρας. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Με το SWIFT, τι θα κάνουμε, ποιος θα λογοδοτήσει. Υπάρχουν ένα σωρό προσφυγές και κοινοποιήσεις από μια σειρά χωρών. Δεν ξέρω, δεν ξέρω είναι η άγρια δύση και πάλι. Αυτό είναι το τοπίο. Από το 1990 το λέμε. Υπήρχαν τέτοιε προοπτικέ και τώρα υπάρχει κυβερνητική δράση σε επίπεδο άγρια δύση. Σαν western. Με το facebook λόγου χάρη. αυτοί που συλλέγουν τα δεδομένα θα γίνουν δισεκατομμυριούχοι έτσι στα γρήγορα και θα κάνουν ό,τι θέλουν τα δεδομένα, δεν ξέρω. Πάντω βλέπουμε ότι μέχρι και το Κογκρέσο έχει φτάσει να νομιμοποιήσει όσα γίνονται. Το είπαμε με την περίπτωση ΦΑΙΖΑ. Ε, η δεύτερη ερώτηση είναι ποιο λογοδοτεί. Στην περίπτωση των ΗΠΑ λόγω χάρη. Για πράγματα που έγιναν ε, ανάρμοστα, α πούμε. Κατά την προσωπική μου άποψη, το χειρότερο που έγινε στην περίπτωση τροπολογία λειτουργία του Φάιζα, και πριν από αυτό βέβαια, είναι ότι οι εταιρείε είχαν ασυλία για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση. Αυτό τους προσφέρθηκε. Και αυτό δεν επέτρεψε καμία νομική προσφυγή την άσκηση κανένα ένομου ε, ένδικου μέσου κατά των εταιριών. Η πολιτεία των κοινωνιών, των κοινωνία των πολιτών δεν μπορούσε να ζητήσει από τι εταιρείε να λογοδοτήσουν βάσει ποια νομική ε, διάταξη έκαναν όσα έκαναν. Πρέπει να πάψει αυτό. Δεν μπορεί να μην λογοδοτούν ποτέ οι εταιρείε. Δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία με τι κυβερνήσει ε, μόνο επειδή του αρέσει η ιδέα. Ε, έτσι ξεκίνησε το SWIFT. Α είμαστε καλοί, α του δώσουμε τα δεδομένα επειδή τα ζήτησαν. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μεταξύ εταιρεών και κυβερνήσεων. Δυστυχώ για την ώρα όμω τα πράγματα έχουν αλλιώ. Διότι το νέο πρότυπο ό,τι αφορά τι σχέσει εταιρεών κυβερνήσεων είναι ότι οι κυβερνήσει λένε στις εταιρείε «Ε, συνεργαστείτε μαζί μα και θα φτιάξουμε ένα ωραίο νομικό καθεστώς με του νόμου μα για να μπορείτε να λειτουργήσετε όπω σας βολεύει. Αν αντισταθείτε δεν θα πάτε πουθενά. Με τι οπτικέ ίνες λόγω χάρη υπάρχουν hacker που μπορούν να αντλήσουν δεδομένα από εκεί. Πώ θα λύσει κανεί το θέμα ε, του PRISM ε, όταν υπάρχουν τέτοια κέντρα hacker. Δεν υπάρχει νόημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό καθεστώ δεσμευτικό, αυστηρό. Σα αρέσει ή όχι, έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώ ζούμε και πάλι σε western. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω μόνο, καθώς βαίνει προς το τέλος αυτή η ενότητα, ότι με την επιφύλαξη των στοιχείων που έχουμε από την Ίνσεν, εμείς δεν έχουμε άμεση πρόσβαση ε, σε στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Και χαίρομαι που είχαμε τον πρώην διευθυντή, ε, τον νομικό διευθυντή και όλα στο MI5 και MI6, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα ε, και πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ τιμή, λοιπόν η συνεισφορά σας και σας ευχαριστώ. Και επίσης και η άποψη της Privacy International είναι άκρος ε, χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Συνεχίζουμε. Μαραθώνια συνεδρίαση σήμερα. 9 η ώρα το πρωί αρχίσαμε, για να καταλάβετε. Δεν φταίω εγώ η γραμματεία, τα παράπονα στη γραμματεία. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν. Τέταρτη ενότητα. Είναι εδώ ο κύριος Πρίμπε. Δεν είναι κύκλισμα των θυρών. Ε, να το γνωρίζετε όσοι θέλετε να ενδιαφέρεστε, δεν είναι και κλεισμένο των θυρών. Είναι ενημέρωση για ε, την ομάδα εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων ε, Πολιτειών. Είναι μια διατλαντική ομάδα αυτή. Συνάδελφοι, παρακαλώ να έχετε πλήρη συνέστηση του χρόνου. Θα πρέπει όλοι να έχουν την ευκαιρία. Αν και οι βασικοί ε, ενδιαφερόμενοι είναι εδώ, μιλάμε για τον πυρήνα της όλης ε, και το, το, το στυλοβάτι της Επιτροπής μας, το στυλοβάτι που είναι μαζί μας από τις 9 το πρωί. Έχουμε και πέντε λεπτά εξοικονόμηση χρόνου. Εδώ θα περάσουμε τώρα να μιλήσουμε για την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτείων διατλαντική ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τελευταίο μέρος της σημερινής ημέρας, απενημέρωση από τον κύριο Νέμιτ, Τώρα δεν θυμάμαι πότε τελευταία φορά συζητήσαμε το θέμα αυτό. Α, χθε μόλι. Ναι, ναι, ναι. Θα σα δώσω το λόγο, απλώ κοιτάζω και το χρόνο. Δεν θέλω να διαμαρτυρηθούν ε, συνάδελφοι. Έχουμε και προσκεκλημένου, όλοι έχουν πτήσει μετά. Ε, και οι άνθρωποι που μένουν εδώ θέλουν να πάνε και σπίτια του. Α είμαστε κάπω ταχεί, γιατί πολλοί έχουν φύγει. Και ε, ο καθένα έχει το τρένο του, αεροπλάνου του να προλάβει. Έχουμε πόσο. Μια ώρα. Ε, δεν το βλέπω έτσι εγώ. Τι σα ρώτησα. Μη λέτε τίποτα. Να ξαναμιλήσετε. Να πάμε γρήγορα λοιπόν. Αυτό είναι το βασικό. Συνέχεια κάθε εδώ πέρα δίπλα μου και μου λέει έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, μην το κάνουμε έτσι και τώρα. Γρήγορα λίγα και κάπως έτσι μια γρήγορη τοποθέτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συναντηθήκαμε και χθε ε, για τρίτη φορά με τα πλαίσια τη αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ. Μια συνάντηση που προβλεπόταν εδώ και δέκα μέρε από την προηγούμενη συνάντησή μα στην Ουάσιγκτον. Όμω, λόγω των πρόσφατων αποκαλύψεων, οι Αμερικανοί ζήτησαν αναβολή. Αυτή ήταν η το, αυτό ήταν το αρχικό πρόγραμμα, αναβλήθηκε τέλο πάντων η συνάντηση αυτή. Ο κύριος Σφάτς από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, και ο κύριος Λί, ο οποίος είναι Γενικός Σύμβουλος της, του Εθνικού Φορέα για την Εσωτερική Ασφαλεία, στο Λευκό Οίκο. Και συντάκτης αλλά και εκδότης όλων των νόμων για τις μυστικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ. Και πάρα πολύ ενεργός και απασχολημένος με τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ. Και την εκπροσώπηση της κυβέρνησης της ΗΠΑ σε ακροάσεις, συνομιλίε, συνεδριάσεις των φορέων εποπτείας. Η χθεσινή μας συζήτηση βασίστηκε σε ένα μακροσκελή κατάλογο με ερωτήσει που κάλυπταν το πεδίο και τους περιορισμούς του τμήματος 7.2 του νόμου Φάιζα. Το ίδιο και για το κεφάλαιο 15, της μεθόδους μεταφοράς δεδομένων προς την κυβέρνηση, τη χρήση των συγκεντρωμένων ή απαιτούμενων δεδομένων, την διάδοση και την τήρηση των δεδομένων, το γεωγραφικό, γεωγραφικό εύρος της συλλογής, τους ποσοτικούς δείκτες για τον αντίκτυπο του προγράμματος τους Ευρωπαίους και ένα ειδικό κεφάλαιο για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες, 1-3-3. Καθώς και το θέμα αν υπάρχουν επιπλέον νομικές βάσεις. Και τέλος, ποια, ποιος ο βαθμός ασφαλείας σε σχέση με, τους, με τις ιδιωτικές εταιρείε που μπορεί να μεταφέρουν πληροφορίες. Σε γενικές γραμμές νομίζω μπορεί να πει κανείς ότι η συζήτηση σε σύγκριση με προηγούμενες συναντήσεις ήταν περισσότερο επικοδομητική. Η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Πριν από τη συνάντηση αυτή τη εβδομάδα, ο Eric Holder, ο Γενικό Αγγελέα των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τι ανησυχίε περί προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων, ε, αναθερώντα τι πρακτικέ ε, τη Αμερικανική κυβέρνηση ε, προ την εποπτεία. Και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, ένα άνοιγμα προ τι μέρημνε των Ευρωπαίων. Ω προ την ατμόσφαιρα λοιπόν των σχέσεών μα, αυτό αντικατοπτρίστηκε και στη χθεσινή συζήτηση. Η Αμερικανική αντιπροσωπεία μας έκανε αντιληπτό το γεγονός ότι τα πράγματα εξελίσσονται χωργά στις ΗΠΑ και η Αμερικανική κυβέρνηση καθώς και το P-Club, ο φορέας δηλαδή που είναι υπεύθυνος για την εποπτεία αλλά και η ομάδα για την αναθεώρηση που συνέστησε ο πρόεδρος Ομπάμα και ο καθηγητής ε, Φάιμπερ είναι ανοιχτή σε προτάσει για το πώς οι αμερικανικοί νόμοι και οι σχετικέ διατάξει θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο συμβατή με τι απαιτήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα. Ο κύριο Λίτ, γενικό Σύμβουλο τη Υπηρεσία, του Διευθυντή για τι μυστικέ υπηρεσίε και την Εποπτεία, ε, μίλησε για τα ειδικά όρια τη συλλογή δεδομένων, για τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων είναι ο κ. Σπέτ, βοηθό του Γενικού Εισαγγελέα και μέλο του Υπουργείου Δικαιοσύνη, επικεντρώθηκε σε θέματα μεταφορά και τήρηση των δεδομένων. Λάβαμε κάποιε χρήσιμε διευκρινήσει, ωστόσο τίποτε που να μην είναι γνωστό δημοσίω τα βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χίδιν συλλογή δεδομένων, τη συλλογή εντός Ευρώπης και τον αριθμό Αμερικανών πολιτών που τους αφορούν όλα αυτά, αυτά παρέμειναν αναπάντητα. Σε κάποια σημεία, επτά σημεία της συζήτησης, η Αμερικανική αντιπροσωπεία επισχέθη να ξαναρωτήσει και να μας πει εάν μπορεί κάτι να γίνει. Μπορεί δηλαδή να μας αποστείλει πρόσθετες πληροφορίες. Ένα παράδειγμα. Βάσει των Αμερικανικών νόμων η Αμερικανική κυβέρνηση υποχρεούται να υποβάλει ετησίως έκθεση για το πώς οι Αμερικανοί πολίτες καλύπτονται, αναφέρονται σε εκθέσεις που συντάσσονται βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από μυστικές υπηρεσίες και μετά ε, τις παραλαμβάνει ο πρόεδρος ή άλλες κυβερνητικές αρχές υπηρεσίες. Ρωτήσαμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε ε, έναν ενδεικτικό αριθμό για το τι γίνεται με τον ανάλογο αριθμό των Ευρωπαίων. Πόσοι αναφέρονται σε τέτοιε εκθέσει εφόσον δημοσιοποιείται ο αριθμό των Αμερικανών. Ίσως τουλάχιστον να μα λέγατε περίπου πόσοι Ευρωπαίοι ε, εξετάζονται. Αυτό είχε να κάνει και με το αρχικό μας ερώτημα. Δηλαδή πόσα ευρωπαϊκά τηλεφωνικά ε, νούμερα ε, καταγράφονται βάσει του άρθρου 15 του Φάιζα πόσα δεδομένα συλλέγονται από, από ευρωπαϊκέ εταιρείε και το καθεξή. Τέλο πάντων, αυτέ οι ερωτήσει παρέμειναν αναπάντητε. Η Ευρωαμερικανική πλευρά επίση μα έκανε μια σύντομη επισκόπηση των συζητήσεων για τι επικείμενε μεταρρυθμίσει στι ΗΠΑ. Εξήγησαν ότι υπάρχουν ε, προτάσει που εξετάζονται για τα δικαιώματα ε, απορρίτου των Αμερικανών πολιτών, των προσώπων. Όμω επίση δήλωσαν ότι υπήρχε μέρημνα για το τι γίνεται με τα δεδομένα των μη Αμερικανών πολιτών και των Ευρωπαίων ειδικότερα η Αμερικανική πλευρά ζήτησε οι Ευρωπαίοι να διορθώσουν πολύ πιο συγκεκριμένα τι απαιτήσει του σχετικά και ήταν καλό που ακούσαμε ότι και από την δική μα αντιπροσωπεία αλλά και από τον Αντιπρόεδρο δηλώθηκε ότι υπάρχει εδώ ένα ένας σημαντικό αντίκτυπο. Ε, αυτό λοιπόν ε, γνωστοποιήθηκε στο P-Club είναι σημαντικό ο κύριο Σφάιερ να το λάβει υπόψη του καθώ θα ενημερωθεί και ο αρμόδιο φορέα εποπτεία. Η Επιτροπή τώρα ετοιμάζει από κοινού με την Προεδρία μια έκθεση, μια κοινή έκθεση που θα υποβληθεί στην Κορεπέρ. Εν ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσει. Κύριε Πίπε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, ωραία. Υπάρχουν ερωτήσει, ε, εάν υπάρχουν ερωτήσει μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. όπω είπατε, μαζί με το P-Club ε, ε, κάναμε μια επισήμανση. Ετοιμάσαμε ένα κείμενο και νομίζω τα μέλη που είναι εδώ είναι και μέλη τη αντιπροσωπή. Θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε πλήρω την Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή την εβδομάδα, θα γίνει στη συνέχεια. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτε. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η συζήτηση και τώρα. Και επίσης υπάρχει και η ομάδα για τις μεταρρυθμίσεις του Πρόεδρου. Νομίζω ο σύμβουλος, όπως είπατε, ήταν χθε στη συνάντηση μαζί σας. Υπήρχαν συγκεκριμένε ερωτήσει. Λοιπόν, με τη σειρά πάλι. Κάρλος, θες να πεις κάτι? Έχεις ερώτηση. Ωραία. Ο Γιάνν. Γιάνν, θες να ρωτήσεις κάτι. Ο Σκιώδης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση. Έχω ένα ερώτημα. Μετά από όλη αυτή τη δουλειά και με βάση αυτά που μας συνοψίσατε, ποιο άλλο βήμα επόμενο μπορεί να πάρει να κάνει η Κομισιόν η η Επιτροπή μας για τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων για την μαζική παρακολούθηση των πολιτών στην Ένωση. Κορνιλία, θέλεις τι να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πάνω κάτω αυτά περίμενα να μας πείτε. Αυτά που ακούσαμε μόλις. Ξέρω ότι μπήκατε σε μεγάλο κόπο και είχατε και προβλήματα και το δέχομαι. Αλλά αριθμό δεν έχουμε για το πόσοι Ευρωπαίοι παρακολουθούνται και φαγγελώνονται. Ωραία, το σημειώνει η Αμερικανική κυβέρνηση ε, αυτές τις ανησυχίες μας. Μπράβο, καλοσύνη τους. Φιλικό το βρίσκω. Εσείς τώρα τι περιμένετε από αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων, τη διατλαντική. Τι μέλη γενέστε. Τελείωσε η υπόθεση μας, τα πάνε. Δεν έχω <laughs> καταλάβει το αντικείμενο και θέλω να προβοκάρω και λίγο με την ερώτηση. Γιατί ξέρετε ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες, αλλά με αυτά που μας είπατε δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Δεν φταίτε εσείς, το ξέρω. Και προφανώς τέτοια απάντηση θα παίρναμε. Αφού η άλλη πλευρά αυτά σου λέει Τη διατλαντικής ομάδα η εταίρα πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες. Έχω λίγο την αίσθηση από τις επαφές που είχαμε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα ότι κατάλαβαν τις ανησυχίες μας ε, και την ανάγκη που έχουμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις για το TTIP, τη συμφωνία αυτή που έχει και πολλά να κάνει με την ψηφιακή πλέον οικονομία και ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό γρήγορα για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε σε αυτή τη συμφωνία. Υπήρξε όμως ένας τομέας όπου η θέση τους ήταν πολύ συμπαγής. Με κάποιες αποχρώσεις, αλλά τα είχαν στυλώσει. Οι δικαστικές αποζημιώσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν πιαστεί σε αυτή τη μέγενη. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν προβλέπεται τέτοιο πράγμα για τους Ευρωπαίους παρόλο που σε ορισμένες υπηρεσίες ε, βρήκαμε ένα ευήκον ους, ε, μας είπαν ότι ναι για πείτε μας να μάθουμε και από τη δική σας εμπειρία τι συμβαίνει. Αλλού όμως σε άλλες υπηρεσίες και σε Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά, στο State Department, τι να πω, πώς να το πω. Ε, μας είπαν ξεχάστε το, αποκλείεται. Γιατί αν το ζητήσουν οι Ευρωπαίοι και τους, ε, το παραχωρήσουμε, θα έρθουν οι Αφγανοί να μας χτυπήσουν την πόρτα. Ναι, άνθρωποι είναι και οι Αφγανοί, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Ε, πώς προχωρούν εκεί οι συζητήσεις, αν προχωρούν. Μπρικίτε Σίπελ, θέλετε να κάνετε ερώτηση εσείς, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. Ακούμε πολλές ε, δηλώσεις, έχουμε πολλές εκθέσεις, πολλές δεσμεύσεις και δύσκολα μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Και μου θυμίζει αυτό μια γερμανική παροιμία που λέει «Καλή εμπιστοσύνη, καλύτερος ο έλεγχος». Και ακριβώς στον έλεγχο όμως δυσκολευόμαστε να βρούμε εκείνους τους μηχανισμούς που προσφέρονται για την εποπτεία. και ρώτησα και από άλλους εμπειρογνώμονες να μάθω πώς θα εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα αλλάξει η κατάσταση. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τον προπολογισμό της NSA. Είναι 700 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δεν με νοιάζει αν είναι ευρώ ή δολάρια. Και η NSA έχει 37.000 υπαλλήλους. Mm. Η NSA και μόνο 37.000 απασχολούμενοι. Κάπως πρέπει να τους απασχολούν. Τι θα κάνουν, θα τους απολύσουν αύριο επειδή εμείς διαφωνούμε. Πώς θα καταλήξουμε σε άλλα αποτελέσματα και με ποιους μηχανισμούς. Και θέλω να προβοκάρω λίγο με την εξή παρατήρηση. Δεν χρειάζεται να απαντήσουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είναι και αρμόδιοι άλλωστε, αλλά διερωτώ με και με βάση αυτά τα πράγματα γιατί δεν τολμούμε και το Συμβούλιο αλλά και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP μέχρι να λυθούν αυτά τα πράγματα για να στείλουμε και κάποια μηνύματα έτσι πιο δυνατά και πιο χειρά. Ευχαριστώ Βρήκητσε. Μια τελευταία ερώτηση από πλευρά μου. Πολ. Ε, χτες πρέπει να σας πω ότι ε, συζητήσαμε με το διευθυντή της NSA στην Ουάσιγκτον και άκουσε και αυτός, ε, ε, ήταν και μέρος της παρουσίασης στο λόφο εκεί του Καπιτολίου και μας είπε Και πώς το αξιολογείτε τώρα αυτό, αυτή την παρουσίαση, είναι, έχουν μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη στρατηγική, ότι να βγαίνουν προς τα έξω τώρα και να ανακοινώνουν και να επικοινωνούν τι κάνουνε. Μετά από μια μακρά περίοδο που έλεγαν ουδέν σχόλιο για θέματα πληροφοριών. Τώρα το έχουν γυρίσει. Ε, ήρθε ο διευθυντής, παρουσίασε τη θέση του. Έχω την αίσθηση ότι είναι προσωρινό αυτό αλλά σχολίαζα και την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μαζική ε, παρακολούθηση και τις κατηγορίες για φακέλωμα. Ποια είναι η στρατηγική, ποια είναι η αίσθησή σας για την Διατλαντική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Θα ασχοληθείτε με περισσότερες καταγγελίες, θα τις σχολιάσετε, γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα τώρα στην επιφάνεια. Γιατί αυτές είναι μάχες που έχουν να κάνουν ε, και με την έρευνα τη δικιά μας και με τις κυβερνήσεις ε, τις ευρωπαϊκές και γενικότερα. Αυτά που μας είπε ο Διευθυντής, δεν ξέρω αν μπορείτε να το σχολιάσετε δημόσια, είναι ενδιαφέροντα ως στρατηγική. Ξέρω ότι ρώτησαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα τελευταίο. Η τελική σας έκθεση πότε θα δημοσιευτεί και πότε είναι και η επόμενη σας συνεδρίαση. Αυτά τα λίγα ερωτήματα. On the question of, um, τα επόμενα βήματα. Νομίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να πούμε ότι το επόμενο βασικό βήμα είναι η έγκριση του κανονισμού. Γιατί η βασική πηγή ενημέρωσης για την NSA είναι οι δυτικές εταιρείε. Και ο κανονισμός είναι πολύ σημαντικός και θα ρυθμίζει ότι ε, μάλλον τι μπορούν να διαβιβάζουν και τι όχι αποδεδομένα οι εταιρείε. Αυτό είναι σαφέστατη προτεραιότητα. Τώρα για την ομάδα εργασία. Η εντολή, το κείμενο που ενέκρινε κορεπέρ δηλαδή, είναι ότι θα αναφέρει η Επιτροπή και μετά θα ληφθούν ε, περαιτέρω αποφάσεις. Λοιπόν, θα πάμε εμεί να αναφέρουμε εκεί και θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Αν θα συνεχίσει τη λειτουργία της ή αν θα διαλυθεί. Προς το παρόν, όπως σας είπα, η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών ε, έφυγε με 7 ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν. Πριν ολοκληρωθεί η έκθεση προς την Προεδρία και ελπίζω πριν τα τέλη του έτους να έρθει αυτή η έκθεση. Το ίδιο ισχύει και για την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς αξιολογεί τα γεγονότα αυτά καθώς επίσης και το θέμα του ασφαλούς λιμένος. Αυτά είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα που έχουμε υπόψη μας. Βέβαια υπάρχει σύνοδος κορυφής δικαιοσύνης και εσωτερικών. 18 Νοεμβρίου θα συναντηθεί με τον Έρικ Χόλτερ, αντιπρόεδρος. Είναι σημαντικό ρώσιμο αυτό. και ποια είναι τα μέσα που πρέπει να εξετάσουμε και να εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η συμφωνία TTIP, αλλά να πούμε ότι όλα αυτά που συζητούμε έχουν να κάνουν και με την, ε, ε, την ε, συνεργασία μας για την ασφάλεια. Έχουμε το TFTP, το PNR, δεδομένα των επιβατών. Έχουμε και άλλες συμφωνίες ασφαλείας με τις Ηνωμένε Πολιτείες και το έχουν καταλάβει. Ότι, οτιδήποτε κάνουμε στη σχέση μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες, είτε αυτό γίνεται βάσει συμφωνιών ή άλλων διευθετήσεων, βασίζεται πάντα στην εμπιστοσύνη. Και είναι σημαντικό να επανέλθει αυτή η αλλων διαφθετησεων βασιζεται παντα στην Είναι οικονομικό θέμα και η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο την εμπιστεύονται οι πολίτες, είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται ή δεν τις χρησιμοποιούν επειδή φοβούνται μήπως τους φακελώσουν και ε, κρατάνε τα δεδομένα τους. Αλλά και γενικότερα για την ε, συνεργασία ασφαλείας χρειάζεται εμπιστοσύνη. Και αν με ρωτάς, Κλοντ, που είναι η νέα στρατηγική ε, διαφάνειας και που το πάει η NSA, έχουν γίνει διάφοροι διάλογοι ε, με την ομάδα επαφής, αντιπρόεδρο και βουλευτές εδώ και κατάλαβαν διάφορα πράγματα. Πρώτον, κατάλαβαν ότι είναι καλή η διαφάνεια, η περισσότερη διαφάνεια, καλή μεν, αλλά δεν αρκεί για να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Καλό είναι να γνωρίζεις ότι σε φακελώνουν γενικώ και αγρίως, αλλά αυτό δεν κάνει τον κόσμο πιο ε, φιλικό προς τα νέα προϊόντα και τα νέα εργαλεία του διαδικτύου. Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογή. η εμβέλεια, τι συλλέγουν, για ποιο λόγο, για ποιους σκοπούς. Και οποιαδήποτε κίνηση που θα φύγει από τα γενικά και τα όριστα και τη μαζική συγκέντρωση χίδιν δεδομένων θα βοηθήσει για την εμπιστοσύνη. Και ένα τρίτο, επίσης δεν είναι αρκετό να ε, μην μιλάμε για το πεδίο εφαρμογής και συλλογής των στοιχείων, απλώς για τη χρήση των δεδομένων μετά. Βοήθησε λοιπόν αυτή η αποστολή να καταλάβουν ότι υπήρχε μια παρανόηση στην αρχή. Ε, θεωρούσαμε ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, όχι ότι τα συλλέγουν. Εντάξει, μωρέ, τα μαζεύουμε. Ενώ για την Ευρώπη, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, η προστασία των πολιτών αρχίζει από τη στιγμή που συλλέγεις τα στοιχεία, όχι τι θα τα κάνεις. Το γεγονό και μόνο ότι τα συλλέγεις. Για τους Αμερικανούς συλλογή στοιχείων είναι μόλις μπει ο αναλυτής και αρχίζει να τα μελετάει. Για μας συλλογή σημαίνει ότι η πρώτη φορά που βάζει χέρι στα δεδομένα είναι ένας κρατικός φορέας. Και ακόμα και αυτή η πρώτη επαφή, η περίφημη ιστορία με τα ε, ε, διατλαντικά, ε, υπερατλαντικά καλώδια, υποβρύχια κτλ. Από εκεί αρχίζει. Και από εκεί και πέρα είναι η χρήση και τα άλλα δικαιώματα, δικαιώμα στην πρόσβαση, στη διαγραφή του, στην απάλληψη και στις δικαστικές αποζημιώσεις. Ε, να πω κάτι τώρα για τις προσφυγές, στις δικαστικές. Ε, αυτό είναι ένα θέμα πολύ παλιό και για τη συμφωνία ε, τη γενικότερη για την ανταλλαγή ε, δεδομένων για την επιβολή του νόμου, όχι τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών. Και ο πρόεδρος το έκανε αυτό. Και τι συμβαίνει σήμερα. Ε, οι Αμερικανοί πολίτες που έρχονται στην Ευρώπη έχουν πλήρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην αποζημίωση γιατί στην Ευρώπη είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ανθρώπινο! Όχι πολιτικό δικαίωμα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, Οποιοςδήποτε έρχεται στην Ευρώπη και ζητάει ασυλό, Αφγανιστάν, Ρωσία, Βόρεια Κορία, δεν ξέρω από πού, ο καθένας έχει το δικαίωμα να το εξετάσει το αίτημά του δικαστής. Από την άλλη, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην προστασία δεδομένων, αλλά και αυτό που συζητούμε τώρα για τη Συμφωνία Ομπρέλα, τη λεγόμενη, προς το παρόν, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο στους Αμερικανούς πολίτες. Και είναι γεγονός ότι ακριβώ αυτό επιζητούμε εμείς, η μεταχείριση για Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό μπορεί να λυθεί στη συμφωνία αυτή, τη συνολική ομπρέλα και ελπίζουμε ότι το έχουν καταλάβει και εκείνοι για να επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ που αναφέρεσε και αυτή στη συνολική συμφωνία ομπρέλα όπως ονομάζεται. Ευχαριστώ, ξέχασα να το ρωτήσω κι εγώ. Κύριε Πρίμπε, θέλετε να πείτε τίποτα πάρα πολύ σύντομα για να τελειώνουμε σιγά σιγά. πολύ σύντομα και για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος. Νομίζω σημαντικό είναι να ξαναϋποθεί ότι είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτών των τριών συναντήσεων ότι πρόοδο έγινε. Ο λόγος που υπήρξε πρόοδος είναι προφανώς πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα ότι καθίσαμε πολλές ώρες μαζί και μιλήσαμε. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνη στην ομάδα. Έπειτα και τα πρόσφατα γεγονότα της κυβέρνησης, της προβλεπόμενης αναθεώρησης, αλλά και αντίδραση της κοινή γνώμης ε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτά που είχαμε ακούσει από το Σεπτέμβριο στο Λουξεμβούργο. Την ακύρωση επίσκεψης Βραζιλιάνου επισήμου στις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου της, της Προέδρου της Βραζιλίας. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Επειδή είδαμε και τις δικές σας αντιδράσεις και ότι υπήρχαν έντονα συναισθήματα σχετικά, όλα αυτά ευαισθητοποίησαν για να γίνουν κάποια περαιτέρω βήματα περί διαφάνειας. Επίσης, το θέμα του κατά πόσο μια νέα στρατηγική ε, NSA μπορεί να προχωρήσει, δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή τόσο αισιόδοξο, αλλά ήταν καλό που επιτέλους ε, θέσαμε τις ερωτήσεις που θέλαμε εδώ και πολύ καιρό στους Αμερικανούς και πήραμε κάποιες απαντήσεις. Βεβαίως, μπορεί κανείς να πάρει ευκολότερα πληροφορίες όταν μιλάει για νομικά πλαίσια πιο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν φτάνουμε σε ζητήματα που θεωρούν ότι είναι δικές τους ε, επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες που μπορεί να επηρεάσουν τη δουλειά τους. Τέλος πάντων, όσο δύσκολα και αν είναι, κάποια πρόοδος επετέχεται ακόμη και στο θέμα των αριθμών για να καταλάβουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Νομίζω μεγαλύτερη ευαισθησία για τις δικές μας τις μέρημνες. Ναι, υπάρχει και ετοιμότητα, προθυμία μάλλον για περισσότερες πληροφορίες από εκείνους προς τα μας, αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι θα γίνει. Αλλά συζητήσαμε πάρα πολύ για τα ένδικα μέσα και νομίζω οι περισσότεροι από τους ομολόγους μας στην αντιπροσωπή καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως κάποιος είπε, νομικίστικες απαντήσεις είναι αναπόφευκτες. Η Βόρεια Κορέα έχει τέτοια δικαιώματα με την Ευρώπη. Θεωρητικά. Όμω κάποιε συζητήσει παρασκηνίου ε, επέτρεψαν να ακουστούν και κάποιε πρωτότυπε ιδέε για το πώ κάποια πρόοδο μπορεί να γίνει. Έγινε αυτό στα πλαίσια του FTTP και του, TN, του PNR. Ε, το αν ε, η δημιουργία θέση ενό ομπούλτσμαν θα μπορούσε να είναι μια πρώτη λύση για να διασφαλιστούν κάποια πρώτα δικαιώματα και των Αμερικανών πολιτών είναι κάποιε πρώτε ιδέε. Εν θερμό. Πρώτη αντίδραση είναι η απόρριψη, αλλά το σκεφτόμαστε όλοι μαζί, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σε ένα βαθμό λοιπόν, νομίζω είναι θετικέ εξελίξει. Για να δούμε και πού υπάρχουν αποκλήσει στι απόψει. Και αυτό υπόθηκε. Είναι ήδη σαφέ. Είναι ήδη σαφές ότι θα χρειαστεί πολλή χρόνο για να καθορίσουμε τι θα πει συλλογή ευθύ εξ αρχή. Για μας το να διαθέτει κανείς δεδομένο είναι ήδη ε, συλλογή δεδομένων. Για εκείνου είναι το να το τηρούν, να το έχουν λάβει και να το τηρούν σε κάποιο αρχείο. Ευχαριστούμε τους κυρίους ε, Νίμιτς και Πίμπερ. Μαραθώνια σημαίνει συνεδρία. Ξεκίνησε στις 9. Ευχαριστώ πραγματικά θερμά όλους τους συναδέλφους που έμειναν στο τέλος και όλο το προσωπικό και τη γραμματεία, όλους μας τους συνεργάτες, πραγματικά από τις μακροσκελέστερες ε, συναντήσεις που έχω συμμετάσχει και προτρέψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήσασταν εδώ από τις 9, πάρα πολύ κράτησε. Ευχαριστώ και τους προτεκλημένου και τη γραμματεία για την διοργάνωση. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα τις ευχαριστίες. Ευχαριστώ όσους έμειναν από τις 9 ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ.